Όσοι δεν γνωρίζουν την αίθουσα, πρέπει να δουν ότι έχουν τα ακουστικά, έχουν τον αριθμό της καμπίνας την οποία θα παρακολουθήσουν την διερμηνία, τη γλώσσα τους, για να είναι πιο ενδιαφέρουσα η συνάντηση. Ε, ακούτε καλά την ελληνική διερμηνία. Η διερμηνία η ελληνική είναι στο κανάλι 7. Ακούτε τη διερμηνία στο κανάλι 7. Τα ελληνικά είναι στο 7. Εγώ είμαι γκλίδα από το ενωμένο Βασίλειο. Ανήκω στην ομάδα των Φρασίνων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα μοιραστούμε την έδρα σήμερα το απόγευμα μεταξύ όλων των συναδέλφων των πολιτικών ομάδων που ασχολούνται εδώ και καιρό με τα θέματα αυτά του ασύλου. Εγώ Ήμουν εισηγήτρια για το Ευρωπαϊκό ε, Γραφείο Προστασίας και ε, Χορήγησης του Ασύλου. Έπρεπε να ψηφίσουμε την προηγούμενη εβδομάδα εξαιτία ε, του ηφαιστείου, όπως ξέρετε, ανετράπη το όλο πρόγραμμα. Δεν ψηφίσαμε. Θα ψηφιστεί η έκθεση στη δεύτερη σύνοδο του Μαΐου. Και Ξέρουμε ότι το γραφείο αυτό θα λειτουργήσει από τη Βαλέτα, από τη Μαλτά. Επίση, είμαι συγγήτρια για την ε, οδηγία των qualification, όπως λέγεται, την οποία έχουμε αρχίσει για τα διάφορα επαγγελματικά προσόντα και τις εξειδικεύσεις. Θα δούμε αν σιγά σιγά υπάρχει μια θετική ανταπόκριση από το Κοινοβούλιο και από το Συμβούλιο. Ξέρουμε ότι κάποιοι θα είναι πιο θετικοί από άλλου. Τέλο πάντων, είμαι εδώ είμαι με διάφορου συναδέλφου, όπω σα είπα, που ασχολούνται με θέματα ασύλου. Θα μοιραστούμε την Προεδρία. Έχουμε μιλήσει για αυτά τα θέματα και με. Μπορούμε να έρθουμε και σε επαφή και με συναδέλφου των Εθνικών Κοινοβουλίων. Πιστεύω ότι αυτό είναι χρήσιμο. Όπως γνωρίζετε για το θέμα αυτό, υπάρχουν διαφορές όσον αφορά το κεκτημένο για τη χορήγηση ασύλου στις διάφορες ε, χώρες μέλη. Κάποιες πιστεύουν ότι υφίστανται πιέσεις, κάποιους άλλους τους αφορά δεδομένου ότι πιστεύουν ότι δεν υπάρχει αρκετή υποστήριξη από άλλα κράτη-μέλη ώστε να εξασφαλιστεί ότι η χορήγηση ασύλου η δική τους ε, δεν θα είναι θέμα μόνο δική τους εκτίθεση. Σήμερα το απόγευμα θα ακούσουμε την ε, συντονιστές του Ακαδημαϊκού Ικτίου, ε, δικαστές, ε, διαφόρους εκπροσώπους, εμπειρογνώμενες, τους οποίους ζητήσαμε να μας πούνε πώς έχει το σύστημα, πώς μπορεί το όλο δίκτυο να βελτιωθεί για να μπορέσουμε να έχουμε ένα αποδοτικό σύστημα το οποίο να μπορεί να παρέχει προστασία στα άτομα τα οποία την χρειάζονται. Σήμερα λοιπόν θα συζητήσουμε για διάφορα θέματα το θέμα αυτού. Η πλήρη μελέτη πιστεύω ότι σε λίγες μέρες, σε λίγες εβδομάδες θα μας εξηγήσει κάποιος συνάδελφος έτοιμη και βεβαίως όταν θα την έχουμε στην ε, ε, διάθεσή μας, θα πρέπει να τη μελετήσουμε, να μην ε, αρκεστούμε σε αυτά τα οποία θα ακούσουμε σήμερα. Θα, έχουμε, θα δώσουμε σε κάθε ομιλητή 8 λεπτά για την παρέμβασή του και μετά θα δώσουμε το λόγο συναδέλφους για να κάνουν παρατηρήσεις, σχόλια, να μας μιλήσουν και οι συνάδελφοι για τις δικές του εθνικές εμπειρίες, να κάνουν ερωτήσεις για να μπορέσουμε να έχουμε ένα πλήρη φάκελο. Όπως βλέπετε είναι ενδελεχής. Έχουμε και τις εθνικές θέσεις ε, κάποιων κρατών μελών για το θέμα αυτό. Χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση θα δώσω τον λόγο στον καθηγητή Φιλίπ Ντεμπρούχερ, καθηγητή στο Ινστιτούτο Ευρωπαϊκών Σπουδών και την Νομική Σχολή του Ελευθέρου Πανεπιστημίου των Βρυξελών, ο οποίος είναι συντονιστής του Ακαδημαϊκού Δικτύου Οδυσσέας. Euh, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι, είμαστε ευγνώμενοι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που μας ανέθεσε να ολοκληρώσουμε αυτή τη μελέτη για το μελλοντικό κοινό σύστημα χορήγησης ασύλου. Γι' αυτό, στα πλαίσια του δικτύου Οδυσσέας, Έχουμε μία ομάδα εμπειρογνωμόνων ε, μέλη, 12 σε πεντε από διαφορετικά κράτη-μέλη. Οι εμπειρογνώμονε προσπάθησαν να κάνουν μία μελέτη η οποία χωρίζεται να χωρίζεται σε τρία μέρη. Στο πρώτο μέλο μα ζητήσει τελικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, παραθέτω, να δούμε ποιοι είναι οι τρόποι και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του κεκτημένου σε θέματα χορήγηση ασύλου από την Κομισιόν. Για το θέμα αυτό Γενικά, θα ήθελα να πω ότι εκφράζουμε τη λύπη σαν διότι οι διάφορες αξιολογήσεις που γίνονται αφορούν τη νομική πτυχή των ε, ε, όλων μέσων που χρησιμοποιούνται παρά στις πολιτικές τους επιπτώσεις. Και βεβαίως εκτιμούμε ότι ο κανονισμός του Βλήνου δεν αξιολογήθηκε σωστά. Απ' την άλλη μεριά θα πρέπει να τονίσουμε ότι έχουν καταβληθεί προσπάθειες από την Επιτροπή, κυρίως σε σχέση με την αξιολόγηση της οδηγίας για τις διαδικασίες ασύλου, για την βελτίωση της αξιολόγησής της, κυρίως χρησιμοποιώντας την μελέτη αντικτύπου για την αξιολόγησή της. Έχουμε λοιπόν να κάνουμε με μια κατάσταση που έχει θετικά και αρνητικά σημεία. Και το θέμα της αξιολόγησης δεν είναι θέμα ευθύνη μόνο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά σε μεγάλο βαθμό και των κρατών μελών, που δεν δέχτηκαν να ακολουθήσουν τις συστάσεις που έκανε σε μία ανακοίνωσή της στι 28 Ιουνίου 2006 η Κομισιόν για τη βελτίωση των μηχανισμών αξιολόγησης. Ελπίζουμε ότι επί αυτού του θέματο, όταν θα τεθεί σε εφαρμογή το νέο άρθρο 70 της Συνθήκης της Λισαβόνας θα μπορέσει να υπάρξει βελτίωση του μηχανισμού αξιολόγησης. Το δεύτερο μέρος της μελέτης μας συνίσταται στην ανάλυση των προτάσεων αναδιατύπωσης της ε, οδηγίας της Επιτροπής, πρώτης Επιτροπής. Και νομίζω ότι μπορώ να πω εξ ονόματο όλων των συναδέλφων ότι κάνουμε θετική εκτίμηση στις προτάσει που υπέβαλε η Κομισιόν Βεβαίως έχουμε έναν ενδιασμό αρχής όσον αφορά την διατήρηση του συστήματος του Βλήνου, που παρά τις κάποιες προβλεπόμενες βελτιώσεις, κατά την άποψή μας θα πρέπει να αναθεωρηθεί εκβαθέων για να μπορέσει να είναι πιο ισχυρή η αρχή της αλληλεγγύης, έτσι όπως προβλέπει το άρθρο 80 της Συνθήκης Λισαβόνου. Και στην έκθεσή μας θα συμπεριλάβουμε διάφορες προτάσεις για αυτό το θέμα, υπό την ευθύνη του συναδέλφου Μανιάνη, ο οποίος δεν μπορεί σήμερα να σας μιλήσει λεπτομεριακά για το θέμα αυτό, δεδομένου ότι δεν προβλέπεται σήμερα στη μισή διάταξη, αλλά είναι κάτι το οποίο δεν θα παραγνωρίσουμε στην τελική μελέτη. Οι προτάσεις αναδιατύπωσης της Κομισιά σε θέματα συνθήκων υποδοχής διαδικασικών ασύλου, χωρίς ασύλου, είναι κάτι το οποίο θα βελτιώσει την εναρμόνιση της πολιτικής ασύλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα της δώσει μεγαλύτερη συνεκτικότητα. Και κατά την άποψή μας λαμβάνει με τον κατάλληλο τρόπο υπόψη των απαιτήσεων όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη Σύμβαση της Γενέβης με την επιφύλαξη κάποιων σημείων τα οποία θα σας αναφέρει η κυρία Ζακουλεβινέτσι, η συνάδελφός μου. Οι συνάδελφοι Ζακ Ζωμότ και Σουζάνα Σαρολέα, Σιλβί Σαρολέα, συγγνώμη, θα επιστήσουν ιδιαίτερως την προσοχή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις ε, θέματα νομικής φύσεως, τα οποία δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο πολιτικών ε, ε, συμβιβασμών με το Συμβούλιο δεδομένου ότι όπως σας λέγω είναι θέματα που αφορούν την νομική πτυχή. Στα πλαίσια αυτή τη ακρόαση μας ζητήθηκε να επιμείνουμε σε οριζόντια θέματα τα οποία τίθενται για το σύνολο των ε, νομικών μέσων και εργαλείων που διαθέτουμε και συζητούμε. Και οι συνάδελφος Ντεμπός και Μπρόνερ θα μας αναφέρουν θέματα που αφορούν την ταυτοποίηση των ιδιαίτερα ευαλώτων ατόμων που ζητούν άτομο και δεύτερον θα κάνουν την αξιολόγησή τους. Τελικά ο Ιβ Καρλιέ θα σας αναφέρει ποια είναι κατά την άποψή μου τα θέματα που μας απασχολούν όσον αφορά τα μέτρα που μπορούν να λάβουν τα κράτη-μέλη πέραν της δεδαφικής τους επικράτειας. Δηλαδή όταν έχουμε να κάνουμε περιπτώσεις παράνομης μετανάστευσης και τις δυνατότητες που έχουμε για τους πρόσφυγες και οι οποίοι είναι αιτούντες άσυλο. Στο τρίτο μέρος της μελέτης κάνουμε προτάσεις για το κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Χορήγησης Ασύλου. Μπορούμε ήδη να θέσουμε το εξής ερώτημα. Μήπως θα πρέπει μακροπρόθεσμα να προβλέψουμε και μια τρίτη φάση για να θεσπίσουμε αυτό το ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου, για να ανταποκριθούμε στον πύχη που τον έθεσε πολύ ψηλά το Συμβούλιο στα πλαίσια του προγράμματος της Στοκχόλμης. Ο Henri Λαμπάι θα σας μιλήσει για κάποια προτάσεις ε, ρεαλιστικές για να κάνουμε πιο συνεκτικό το όλο θέμα και από τις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής αυτής υπηρεσίας υποστήριξης του ασύλου και λαμβάνοντας υπόψη και τις ε, αποφάσεις και την αρμοδιότητα του Ευρωπαϊκού Δικαστήριου. Κύριε Πρόεδρε, τελειώνοντας θέλω να σας πω ότι με μεγάλη τιμή σας παρουσιάζουμε τα πρώτα πορίσματα της μελέτης την οποία κάναμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Να σας πούμε ότι εκφράζουμε την ελπίδα ότι θα είναι η μελέτη αυτή χρήσιμη και θα ήθελα να προσθέσω ε, προς τους εισηγητές ότι θα είμαστε στη διάθεσή σας κυρίες και κύριοι για να σας βοηθήσουμε στη δουλειά σας που ξέρουμε ότι από πολιτικής πλευράς είναι δύσκολη αλλά εξίσου δύσκολη και από τεχνικής. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Thank you very much for that, um, that introduction to tell us... Ευχαριστώ για την εισαγωγή σας. Μα είπατε ποια είναι τα κύρια σημεία και τα κύρια θέματα που θα ρωτήσετε οι συναδελφοί σα. Και βεβαίω οι συγγητές μα θα είναι σε επαφή μαζί σας. Νομίζω ότι μπορούμε να το καταστήσουμε αυτό ευθύ αρχή απόλυτα σαφέ. Περνάμε στο επόμενο ε, θέμα με τον Ζακ Ζωμότ που θα μας μιλήσει για τις Γενικές Αρχές του Ευρωπαϊκού Δικαίου ως κατευθυντήρες γραμμές για τον ορισμό των δικονομικών εγγυήσεων για του ετούντε άσυλο. Ζακ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κύριοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι. Μου ζητήθηκε εντό λίγων λεπτών να σας παρουσιάσω το θέμα αυτό και σκέφτηκα να παρουσιάσω τις Γενικές Αρχές του Ευρωπαϊκού Δικαίου πρώτα για να φανούν οι συνέπειες, της δικονομικές εγγύησεις για τις διαδικασίες ασύλου. Πρέπει κανείς να έχει υπόψη ότι στη σημερινή εκδοχή της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την για που αφορά τις ε, διαδικασίες ασύλου υπάρχει μια ενιαία διαδικασία για το, καθεστώς, το επικουρικό καθεστώς προστασίας αλλά διατηρείται η αρμοδιότητα των κρατών ε, μελών ε, για την ε, ενίσχυση των ελάχιστων κριτηρίων που προβλέπονται στην οδηγία για τις διαδικασίες ασύλου. Κάθε εθνικό κράτος λοιπόν θα πρέπει να προβλέψει κάτι ανάλογο στην εθνική του νομοθεσία. Η παθή σκοπιά πρέπει να καθοριστεί βάσει ποιων κριτηρίων θα προβλεφθούν κοινέ διαδικασίες μεταξύ των κρατών των ενδιαφερομένων και τι δικαστικές δυνατότητες υπάρχουν εδώ. Ευθύς εξ αρχής ένας προβληματισμός μας ήταν οι νομικές προδιαγραφές που θα επιτρέψουν να δημιουργηθούν κοινέ διαδικασίε και αντιμετωπίσαμε διαφορετικά προβλήματα, όπω η Σύμβαση τη Γενέβη και το πρωτοκολλό τη, που ομόφωνα θεωρείται ότι δεν δημιουργεί δικονομικέ εγγυήσει αυτέ καθεαυτέ. Έπειτα Υπήρχαν ε, και τα συμπεράσματα για τους ε, πρόσφυγες από τον ΟΗΕ που ούτε αυτά προβλέπουν ε, συγκεκριμένα συγκεκριμένες εγγύσεις. Η δεύτερη πηγή που αναζητήσαμε ήταν η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τη διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, αλλά γνωρίζουμε μετά την απόφαση Μαγιού για κι άλλες ότι δεν προβλέπονται συγκεκριμένα κριτήρια. Υπάρχουν και συστάσεις των διαφόρων οργάνων του Συμβουλίου της Ευρώπης, αλλά καμία δεν έχει υποχρεωτική ισχύ. Υπάρχει όμως και η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και τα άρθρα 2 και 3. Συμβάσεις που περιλαμβάνονται και σε το επίπεδο της επικουρικής προστασίας για τα θέματα ασύλου, καθώς και τα όσα προκύπτουν από το άρθρο 13, για το, από το άρθρο 13 για τα ελάχιστα κριτήρια στην περίπτωση του ασύλου. Υπάρχει και μια τρίτη πηγή, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εδώ υπάρχουν δύο δυνατότητες. Πρώτα απ' όλα το άρθρο 47 της Χάρτας των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων που από τη στιγμή που τέθηκε σε, σε ισχύ εγγυάται την δικονομική προστασία για τα υποχρεώσει και τα δικαιώματα των πολιτών της Ένωση και συμπεριλαμβάνει έναν αριθμό ελάχιστων κριτηρίων. Επίσης θα μπορούσαμε να αναφέρουμε για τις διοικητικέ διαδικασίες το άρθρο 41 της Χάρτας που ορίζει τα όργανα, τα σώματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους και θα έπρεπε εδώ να αναφέρουμε και το πώς η οδηγία για τις διαδικασίες εφαρμόστηκε και κατά πόσον ε, εξελέγχθη από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Εδώ όμω δεν υπάρχει συγκεκριμένη νομολογία από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την ε, εφαρμογή, την υλοποίηση τη οδηγία αυτή. Και αυτό εξηγείται ίσω από το γεγονό ότι μέχρι την θέση σε ισχύ τη συνθήκη τη Λισαβόνα οι διαδικασίε και τα προδικαστικά ερωτήματα δεν ήταν ε, δημοσιοποιημένα και δεν ήταν στην δικαιοδοσία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Σε ό,τι αφορά την ίδια την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, όπω και σε άλλα θέματα που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι αποφάσεις που έχει εκδώσει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν αρχές που θα έπρεπε να προβλέπουν αποδοτικές και αποτελεσματικές διαδικασίες στο διοικητικό επίπεδο, ιδίως για την προσφυγή σε μια δικαιοδοσία υπό την έννοια της συνθήκης. Όλα αυτά όμως πρέπει να τα δούμε με ιδιαίτερη σύνεση, γιατί κάθε φορά πρέπει να καθοριστεί εάν πρόκειται για οριζόντια κριτήρια ή ξεδικευμένα ανάλογα με την κάθε υπόθεση. Το πρώτο μας λοιπόν συμπέρασμα είναι ότι δεν έχουμε συγκεκριμένες ε, ειδικέ αρχές πέρα από τις γενικές του Ευρωπαϊκού Δικαίου για το θέμα αυτό όπως προκύπτουν από την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων από τη μια και από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την άλλη. Αυτό λοιπόν που κάναμε σε μια δεύτερη φάση στην ομάδα που ανέλαβε την εξετάση του θέματος αυτού είναι να ορίσουμε βάσει της νομολογίας αυτού του δικαστηρίου έναν κατάλογο, ένα κατάλογο με αρχές, αρχές τις οποίες θα μπορούσαμε να ονομάσουμε γενικόλογες και οι οποίες θα μπορούσαν να καλύπτουν τις δικονομικές εγγύησεις υπό την έννοια της διεθνούς προστασίας. Μία μελέτη αρκετά αμφιλεγόμενη, διότι η Ερμηνεία της, των αποφάσεων του δικαστηρίου είναι σχετική. Κάποιες φορές ε, τα, οι αποφάσεις αφορούν τη συγκεκριμένη υπόθεση. Έπρεπε όμως να δούμε πώς εφαρμόζεται η ισχύουσα οδηγία και τι πρόοδος θα μπορούσε να επιτελεστεί βάσει των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα δώσω λοιπόν τώρα το λόγο στην κυρία Σαρολέα για να σας δώσω δύο συγκεκριμένα παραδείγματα του τι μπορέσαμε να κάνουμε, γιατί όλε τι προβληματικέ μα δεν μπορούμε να σα τι παρουσιάσουμε. Θα σα πούμε λοιπόν δύο συγκεκριμένε περιπτώσει για να δούμε και σε τι συμπεράσματα μπορούμε να καταλήξουμε μια τέτοια προσέγγιση. Voilà, Εντάξει, λειτουργεί. Όπω είπε και ο κύριο Ζωμότ, δύο συγκεκριμένα παραδείγματα, γιατί με το χρόνο που έχουμε εδώ δεν ήταν δυνατόν να κάνουμε μια επισκόπηση όλων των ζητημάτων που προκύπτουν από το τωρινό κείμενο και όλε τι προτάσει. Δύο παραδείγματα λοιπόν. Το πρώτο, το πρώτο που απεικονίζει αυτή τη δυσκολία είναι το δικαίωμα στην ε, νομική αρρωγή, την ε, δωρεάν νομική αρρωγή. Η πρόταση τη τροποποιημένη οδηγία διευρύνει το δικαίωμα τη δωρεάν συνδρομή και για του ετούντε άσυλο. Υπάρχουν κάποιοι κανόνε για την πρόσφαση, βέβαια, για την πρόσβαση, που ισχύουν στην πρώτη φάση τη διαδικασία, στη διοικητική φάση. Εδώ το ερώτημα που τίθεται είναι αν είναι σκόπιμο κάτι τέτοιο και αν μπορεί να είναι και υποχρεωτικό. Η διεθνή δικαιοδοσία λοιπόν θα πρέπει να δούμε αν κάνει αυτή τη διεύρυνση των δικαιωμάτων ε, υποχρεωτική. Δεν υπάρχει για την ώρα σαφή απάντηση, όμω θα μπορούσαμε από την ομολογία να συμπεράνουμε ότι όπω και ο Ζακ Ζωμότα ανέφερε από τι διάφορε αποφάσει κάποιε φορέ για άτομα τα οποία είναι ιδιαίτερα ευάλωτα και για κινδύνου σοβαρού όπω την παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, εκεί είναι ευκταίο και η δικαιοδοσία θα έπρεπε να προβλέψει την υποχρεωτικότητα τη νομικής αρρωγής, της δωρεάν νομική αρρωγή. Το δεύτερο ερώτημα που προκύπτει ένα ερώτημα που συζητάται ιδιαίτερο σε όλα τα εθνικά κρατημέλη είναι το κατά πόσον θα μπορούσε να έχει ανασταλτικό χαρακτήρα η προσφυγή ενό ετούντα άσυλο. Ε, και μάλιστα σε σχέση με μια απόφαση για απομάκρυνση από την επικράτεια. Εδώ θα μπορούσαμε να σκεφτούμε, και πρέπει βεβαίω να είμαστε συνετοί, αλλά αυτή είναι η τάση που προκύπτει από την ομολογία και από τι διάφορε προτάσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή άλλωστε. Όπω τα όργανα που συζητούμε σήμερα, μια πρόσφυγη δεν, μπορού, δεν μπορεί να θεωρηθεί πραγματική παρά μόνο να στέλνει ένα μέτρο από, για την απομάκρυνση από την επικράτεια. Το Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την απομάκρυνση από την επικράτεια το λέει αυτό ξεκάθαρα αυτή τη στιγμή. Όχι απαραίτητο στα θέματα ασύλου, διότι δεν υπάρχουν αναγκαστικά αποφάσει που αφορούν το συγκεκριμένο ζήτημα. Όμω, ο συσχετισμό μεταξύ των δύο ε, νομικών προβλημάτων είναι προφανή. Θα μπορούσαμε λοιπόν σήμερα να πούμε ότι η υποχρέωση αυτή για την αναγνώριση των ασταλτικού χαρακτήρα τη προσφυγή και για να είναι και πραγματική προσφυγή μπορούμε να συμπεράνουμε ότι θα πρέπει να είναι υποχρεωτική αυτή η εφαρμογή και στα ζητήματα ασύλου. Θα παραμένω σε αυτά τα δύο παραδείγματα για να μην ξεπεράσω το χρόνο που μα έχει διατεθεί και φαντάζομαι ότι στη διάρκεια τη συζήτηση θα επανέλθουμε και σε αυτά. Σα ευχαριστώ. Oh, thank you. I mean, those are... Ευχαριστούμε. Αυτά τα δύο ζητήματα που θέσατε είναι ζητήματα που θα προκαλέσουν σίγουρα συζήτηση από το σώμα και βεβαίως ε, και στα εθνικά κοινοβούλια. Είναι λοιπόν να ενδιαφέρον να βλέπουμε θέματα που ούτως ή άλλως θα διερευνηθούν. Τελευταίος ομιλητής για αυτό το τμήμα της συζήτησης είναι ο κύριος Μαγιάννη, στον οποίο ζητήσαμε να απαντήσει στο ερώτημα αν τα κράτη-μέλη μπορούν να εμπιστεύονται το ένα, τα συστήματα ασύλου των υπολείπων. Έχει έρθει κοντά μας ο κ. Μαγιάννη σε πολλές περιπτώσεις Και ήθελα απλώ να δούμε κατά πόσο δεν, αν δεν υπάρχει αρκετή εμπιστοσύνη, τι μπορεί αυτό να σημαίνει για του πολίτε. Θέλουμε λοιπόν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον να ακούσουμε, Φραντσέσκο. Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωκοινοβουλίου, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, είναι πραγματικά μεγάλη τιμή για μένα να μπορώ να σας προσφωνήσω. Να προσφωνήσω τόσο εξέχουσε προσωπικότητες ο συντονιστής του εγχειρήματο Φιλίπ, υπενθύμησε ότι ο χρόνος πιέζει. Θα μπορέσω μόνο να καλύψω ένα από τα θέματα που αφορά το σύστημα του Δουβλίνου και άλλα θέματα καλύπτονται στην έκθεση βέβαια. Ωστόσο με ιδιαίτερη χαρά να απαντήσω ερωτήσεις αν υπάρξουν κάποιες ερωτήσεις και το επιτρέπει ο χρόνος να τεθούν. Όπως η κυρία Λαμπέρ υπενθύμησε, η παρουσίασή μου <clears throat> επικεντρώνεται σε ένα θέμα της συνθήκης πολιτικά Μπορούν τα κράτη-μέλη να εμπιστεύονται σε σχέση με τους ετούντες άσυλο της διαδικασίας. Σε πρωτού προχωρήσουμε είναι αναγκαίο να αποσαφηνίσουμε τι σημαίνει εμπιστοσύνη σε αυτό το πλαίσιο. Με εμπιστοσύνη εννοούμε γενικά ότι θα υπάρχει εμπιστοσύνη ότι ο ετών άσυλο δεν θα κινδυνεύει όταν θα μεταφέρεται σε μια, από, μια, από ένα κράτος μέλος σε ένα υπεύθυνο άλλο κράτος όσον αφορά ταπεινωτική μεταχείριση ή όσον αφορά βασανιστήρια ή μεταχείριση. Εμπιστοσύνη λοιπόν σημαίνει εμπιστοσύνη στο γεγονός ότι η μεταφορά με βάση τις συμφωνίες αυτές θα είναι σύμφωνη με τις αρχές του νομβεφουλμό και έτσι θα μπορεί να λειτουργήσει. Αυτή είναι η νομική έννοια του όρου εμπιστοσύνη σε αυτό το πλαίσιο. Και πάλι μέσα σε αυτό το πλαίσιο ίσως αξίζει να τονίσουμε κάτι. Ότι ο απόλυτος σεβασμός για τον νομβεφουλμό είναι ο ακρογωνιός λίθος ε, επί του οποίου θέλουμε να οικοδομήσουμε το κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου. Επίσης αξίζει να υπο υπογραμμίσουμε ότι ως θέμα διεθνούς δικαίου τα κράτη-μέλη έχουν την υποχρέωση να σέβονται αυτή την αρχή οποτεδήποτε και πάντοτε, ακόμα και όταν έχουμε μεταφορά μέσα σε ένα άλλο κράτος μέλος ε, ενός ετούντος άσυλο. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ήταν σαφέστατο επί του σημείου αυτού, τονίζοντας ότι τα κράτη-μέλη δεν επιτρέπεται να βασίζονται αυτόματα στις ε, συμφωνίες ε, της, του κανονισμού του Δουβλίνου. <clears throat> Και το γεγονός ότι αντί ενός άλλου κράτους, ε, ένα άλλο κράτος μέλος ε, θα έχει ευθύνη εξέταση της αίτηση ασύλου, <clears throat> δεν θα σημαίνει ότι υπάρχει μετάθεση αρμοδιότητας μέσα στο πλαίσιο του νόμου refoulement Μέσα σε αυτό το προήμιο λοιπόν μπορώ προετοιμάζοντας, προλυαίνοντας το έδαφος να έρθω στο κύριο ερώτημα. Μπορούν τα κράτη-μέλη να εμπιστεύονται το ένα το άλλο όσον αφορά το σύστημα ασύλου που έχει εξεταστεί μέχρι τώρα. Λοιπόν, η απάντηση μέχρι τώρα υπό την Σύμβαση της Γενέβης και υπό την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου είναι ότι θα υπάρχει συγκεκριμένη εμπιστοσύνη, όχι απόλυτη ή τυφλή εμπιστοσύνη. Τι είναι συγκεκριμένη, εύλογη εμπιστοσύνη. Αφενός όλα τα κράτη-μέλη είναι συμβαλόμενα μέρη στην ε, σύμβαση της Γενέβης, στη συνθήκη της Γενέβης και στη σύμβαση ε, των ευρωπαϊκών δικαιωμάτων. Και έτσι βασιζόμαστε στο ότι αυτό είναι εύλογη εμπιστοσύνη. Από την άλλη πλευρά είναι σαφές ε, όσον αφορά την διεθνή νομολογία ότι η δυνατότητα πρέπει να υφίσταται ώστε αυτή η αρχή να μπορεί να ε, αντιμετωπιστεί εύλογα. Δηλαδή να αποφεύγει ένα κράτος μέλος ε, όσον αφορά την μεταφορά ενός ετούντος ε, άσυλο από ένα κράτος μέλος σε άλλο, εάν το επίπεδο προστασίας για αυτό το άτομο του ετούντο άσυλο σε ένα άλλο κράτο μέλο θα βρίσκεται κάτω ενό συγκεκριμένου επίπεδου. Αυτή η υποχρέωση να μην μεταφέρεται κάποιο ε, υπό αυτού του όρου. υφίσταται σήμερα. Είναι η ρήτρα sovereign clause, η ρήτρα κυριαρχία. Μπορεί ένα κράτο όταν έχει τέτοιε πληροφορίε να μην μεταφέρει ένα ετούντα άσυλο σε ένα άλλο κράτο μέλο και να εξετάσει την αίτηση ασύλου του το ίδιο. Όπω ελπίζω να έχω καταστήσει σαφέ ε, μέχρι τώρα, αυτό δεν είναι απλά και μόνο μια κατά το ε, ρήτρα. Είναι μια θεμελιώδης ρήτρα ώστε να μπορεί να λειτουργεί το σύστημα με βάση τις ε, διεθνείς ρήτρες για την προστασία των ετούντων ασύλων, ασύλου. Αυτό το θέμα ως ε, θέμα εφαρμογής δικαίου. ως έχουν όμως τα, πράγμα, τα πράγματα σήμερα, αυτή η εγγύηση είναι τόσο σημαντική που η σημασία αυτής της ρήτρας δεν μπορεί να υπερεκτιμηθεί. Όλοι γνωρίζουμε ότι διαφέρουν από κράτος σε κράτος ε, οι προδιαγραφές για τις διεργασίες ασύλου. Και επίσης γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την άποψη της ΥΠΑ της Αρμοστίας των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες, κάποιες τέτοιες προδιαγραφές δεν ευθυγραμμίζονται απόλυτα σε σχέση με τις διεθνείς προδιαγραφές. Έτσι λοιπόν αυτή η ρήτρα είναι πάρα πολύ σημαντική και στη θεωρία και στην πρακτική σήμερα και η ε, ρήτρα <clears throat> κυριαρχία sovereignty clause θα πρέπει κάπως και να ενισχυθεί κιόλα γιατί δεν είναι επαρκή πλήρω. Η πρόταση λοιπόν σε σχέση με την ε, τροποποίηση του συστήματος ε, της, του κανονισμού των διεργασιών Βλίνου θα πρέπει να επανεξεταστούν διότι σε σχέση με την κέρια σημασία αυτών των διατάξεων όπως η πραγματική δηλαδή αντιστάθμιση έναντι των διεργασιών αυτών έχει μεγάλη σημασία. Αυτό σε σχέση με το άμεσο μέλλον. Τι θα γίνει τώρα μακροπρόθεσμα. Θα είναι δυνατόν όταν θα έχουμε μια, ένα κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου να καθορίσουμε ένα κανόνα απόλυτης εμπιστοσύνης. Με άλλα λόγια, θα είναι δυνατόν <clears throat> να άρουμε ένα κανόνα όπως την ρήτρα κυριαρχίας και να υπάρχει η δυνατότητα με βάση ε, ε, λόγους non-refoulement να αμφισβητηθούν οι διεργασίες Δουβλίνου. Εγώ θα έλεγα τουλάχιστον όχι αν το κοινό σύστημα ασύλου αναπτυχθεί με βάση τις ε, σημερινές γραμμές. Επιτρέψτε μου σε αυτό το σημείο τώρα να οδηγηθώ στο, στην κατακλίδα. Αν αναπτυχθεί ένα τέτοιο κοινό σύστημα ασύλου με βάση τις σημερινές γραμμές θα έχει δύο χαρακτηριστικά δομικά που θα είναι σημαντικά. Πρώτον, η υποδοχή των ετούντων άσυλο και η κρίση της αίτησή τους, η αξιολόγησή της θα είναι θέμα των κρατών μελών υπό το εναρμονισμένο νομικό πλαίσιο φυσικά. Δεύτερον, μέσα στο πλαίσιο διεθνούς δικαίου, οι ατομικές ε, ευθύνες και τα καθήκοντα των κρατών μελών θα παραμένουν όπως έχουν σήμερα καταρχήν. Υπό το φως λοιπόν αυτών των δύο χαρακτηριστικών στοιχείων, αν είναι σήμερα η ρήτρα κυριαρχία sovereignty clause, clause μια αναγκαιότητα, θα έλεγα ότι και στο μέλλον θα παραμείνει μια νομική αναγκαιότητα αντί διαδιατάγματος να θεσπίζουμε την ύπαρξη και την επιβολή της απόλυτης εμπιστοσύνης να δράσουμε με βάση αυτή την προσέγγιση. Η εμπιστοσύνη πρέπει και μπορεί να οικοδομηθεί βήμα προς βήμα μέσα σε ένα ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου οι προποθέσει για αυτήν την εμπιστοσύνη πρέπει να ενισχυθούν. Να ευθυγραμμιζόμαστε απόλυτα με το διεθνέ δίκαιο. Να υπάρχουν επαρκεί εγγυήσει ότι όλα τα δικαιώματα θα είναι απόλυτα σεβαστά. Και να υπάρχει δυνατότητα εποπτεία ε, επιμερισμού καθηκόντων και όταν όλα αυτά θα μπορέσουν να λειτουργήσουν σωστά, η δυνατότητα να αμφισβητηθούν οι μεταφορέ αυτέ πάλι θα πρέπει να παραμένει για νομικού λόγου. Όμω η πρακτική τη σημασία και η επίπτωση όσον αφορά την ε, ε, ομαλή η συνεργασία δεν θα έχει πια τέτοια σημασία. Ευχαριστώ. Thank Σας ευχαριστούμε και ευχαριστούμε όλους τους ομιλητές διότι αρχίζουν να καθορίζουν το πλαίσιο των διεργασιών δίνοντας ε, συγκεκριμένα χειροπιαστά θέματα και ερωτήματα τα οποία θα πρέπει να μας απασχολήσουν ώστε να δούμε τι θα μπορέσει να γίνει σε σχέση με το κεκτημένο και όσον αφορά το άσυλο και το θέμα της εμπιστοσύνης είναι ένα θέμα στο οποίο σίγουρα θα επανέλθουμε και στο μέλλον. Γνωρίζω ότι υπάρχουν κάποιοι που θέλουν ίσως ήδη είτε να παρέμβουν κάνοντας κάποια σχόλια σύντομα ή να διατυπώσουν κάποιες ερωτήσεις αλλά δύο λεπτά ο καθένας παρακαλώ για να καταφέρουμε το δυνατόν περισσότεροι να συμμετάσχουν. Θα ήθελα να καλωσορίσουμε από την ε, γερουσία της Τσεχίας τον κύριο Τόμας Κρούζεκ παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα σύντομα να σας ενημερώσω για το πώς το σύστημα του πακέτου ασύλου αντιμετωπίζεται από την Δημοκρατία της Τσεχίας. Η Γερουσία ασχολήθηκε με όλες τις προτάσεις και υπέβαλε γνωμοδότηση από πλευρά τη. Η τσεχική γερουσία συμφωνεί υπερ, ο περαιτέρω εναρμονισμός ότι είναι αναγκαίος στο μέλλον. Από την άλλη πλευρά η γερουσία στην Τσεχία είπε ότι σε κάποιες ε, οδηγίες υπήρχε πολύ λίγο χρονικό διάστημα μεταξύ της εφαρμογής και των νέων προτάσεων. Η Γερουσία λοιπόν δεν πίστηκε απόλυτα ότι υπήρχε επαρκής χρόνος ώστε όλα τα προβλήματα να εντοπιστούν και να αναλυθούν. Όλες οι προτάσεις πρέπει να είναι πλήρεις ώστε να μην χρειάζεται στη συνέχεια αναπροσαρμογή. Και δεν συνιστά η γερουσία οι ετούντες άσυλο να έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Διότι αυτό το μέσο πολλές φορές την χάνει αντικείμενο κατάχρησης. Προέρχονται, έρχονται για οικονομικούς λόγους πολλές φορές στις χώρες μας αυτά τα άτομα και παρακάμπτουν τους κανόνες, που οι κανόνες, ε, τους κανόνες για την μετανάστευση. Και έτσι έχουμε και κάποιες επιφυλάξεις εμείς όσον αφορά την τροποποίηση των κανόνων του συστήματος του Δουβλίνου. Δεν θεωρούμε ότι οι κανόνες αυτοί πρέπει να τροποποιηθούν. Δεν πρέπει να αλλοιωθούν και με βάση οποιαδήποτε, οποιοδήποτε πρόσχημα. Δεν θα πρέπει οι, τα κράτη-μέλη να αρχίσουν να αλλάζουν, να παραλλάσσουν τους κανόνες ώστε να μην υπάρχει, ας το πω έτσι, ενασχόληση με αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Ήθελα να ακούσουμε τη διαρμηνία πρώτα και γι' αυτό καθυστερήσαμε λίγο. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε για την πληροφορία που μας δώσατε για την τσεχική γερουσία σε κάποια θέματα. Και το Δουβλίνο και αυτό το θέμα που αναφέρατε για τον χρόνο. Πόσο χρόνο έχουν τα κράτη-μέλη ώστε να αρχίσουν πραγματικά να δημιουργούν ένα σύστημα το οποίο θα είναι λειτουργικό. Αυτό σίγουρα είναι ένα θέμα το οποίο έχει τεθεί οπωσδήποτε. Η Ελέν Φλότρο παρακαλώ από την Ευρωβουλή. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να επιβληθώ από την ε, παρουσία των ομομαθών εμπεργονομών για να τους κάνω μία ερώτηση για τις ε, επιπτώσεις που προβλέψουν τα υπάρξη από την ε, πρόσβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και κυρίως όσον αφορά τις ε, νομικές διεθνείς μας υποχρεώσεις, όπως αναφέρεται και στην ε, νομολογία, και δεύτερον για το δικαίωμα προσφυγής που θα μπορούσε να συνεπάγεται η επικύρωση αυτής της σύμβασης. Και στον τελευταίο παρεμβαίνοντα μια ερώτηση για τις προοπτικές ενός ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου πιο ισχυρού και πιο κινητοκοκιοποιημένο σε περίπτωση που υπάρχει άρνηση χορήγηση ασύλου από μια χώρα δεν θα ήταν καλό να ρωτηθούμε εάν δεν θα έπρεπε να υπάρχει ένα ευρωπαϊκό δικαστήριο ειδικό για τέτοιου είδους θέματα, για να επιλύει τέτοιου είδους θέματα και να μπορεί κατά κάποιο τρόπο να βλέπει πώς έχουν οι αποφάσεις των εθνικών δικαστηρίων για τέτοιου είδους θέματα και να ενεργεί σε περίπτωση που υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Οι πρόσωποι των Εθνικών Κοινοβουλίων, παρακαλώ, εάν θέλετε να κάνετε ερωτήσεις, είστε ελεύθεροι. Σας καλώ να μην ε, αισθάνεστε ότι μόνο οι ε, Ευρωπαίοι συναδελφοί σας θα κάνω ερωτήσεις. Η Σοφή. Το πρώτο θέμα που ήθελα να θίξω είναι το εξής. Το θέμα της ε, πραγματικής προσφυγής και της νομικής δωρεάν αρρωγής. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ χρήσιμο. Επίσης, εφόσον αυτά εν μέρει απαντήθηκαν ποια είναι, ποιος είναι ο ορισμός, η έννοια της ασφαλής, η σίγουρης τρίτης ε, χώρας. Τι σημαίνει αυτό από άποψη διαδικασίας. Και να ανακαταλείψουμε την ε, ιδέα του ευρωπαϊκού καταλόγου εξαιτίας προβλημάτων που υπήρχαν, αυτή την ε, αναφορά, αυτή η ε, έννοια στην οδηγία, στο κείμενο της οδηγίας θα πρέπει να συνεχίσουμε να την έχουμε ή στο παράρτημα 2 να ε, κάνουμε κάποια αλλαγή όσον αφορά τον κατάλογο τρίτων χωρών ασφαλών όσον αφορά τη χώρα προέλευσης του ετούντος άσυλ. Επίσης, κάτι να μου πείτε για την έννοια της ευρωπαϊκής χώρας σίγουρης, της ασφαλούς. Δεδομένου ότι το θέμα αυτό κατά την άποψή μου τώρα δεν έχει λόγο ύπαρξης και χρησιμοποιείται πολύ λίγο. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε αν αυτή η έννοια ή μάλλον ποιο είναι το μέλλον της, τι προβλέπετε για την έννοια αυτή στα νέα κείμενα και την άποψή σα. Και κάτι που θα σας φανεί παράξ στην ε, συνεδρίαση των σκιωδών εισηγητών του θέσαμε το ερώτημα χωρίς να δώσουμε οριστική απάντηση. Αναρωτηθήκαμε λοιπόν από ποια στιγμή ένα άτομο μπορεί να θεωρηθεί ως τον άσυλο στην πραγματικότητα. Διότι η χρονική προθεσμία των 72 ωρών που προβλέπεται από τη στιγμή που κάποιος καταθέτει επισήμω την αίτηση ασύλου ε, μετράει ο χρόνος. Πώς ακριβώς μετράει για να μπορέσουμε να το καθορίσουμε αυτό με σαφήνεια. Ευχαριστώ εύκολα. Κάποια εύκολα ερωτήματα από ό,τι φαίνεται. Θα θέλαμε να δώσουμε κάποια συνέχεια σε αυτά. Παρακαλώ. Ο ρόλο μου είναι πολύ απλό. Αν επιτρέπετε για το πρώτο ερώτημα, θα ήθελα να σα προτείνω την ερώτηση να την αναβάλουμε γιατί την στιγμή κατά την οποία ο Ρίλα Μπέλ θα κάνει την του, διότι πιστεύω ότι θα σας απαντήσει πράγμα που θα μας επιτρέψει τώρα να κερδίσουμε χρόνο δεδομένου ότι έχουμε μόνο λίγα λεπτά στη διάθεσή για πάνω στις ερωτήσεις. Αντιθέτως, για τα προβλήματα και τα θέματα διαδικασίας θα απευθυνθώ στους συναδέλφους Ζωμότ και Σαρολέα. Πάρα πολύ σύντομα θα επανέλθω στο θέμα αυτό το οποίο μου ζητήσετε, αν συγκρίνει κανείς την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, δεν μπορούμε να πούμε ότι γενικά η έννοια στην ομολογία αυτή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων η... όταν ένα δικαίωμα σταματά να χορηγείται είναι κάτι το οποίο βρίσκουμε με σαφήνεια. Όταν κάτι τέτοιο ε, ένα τέτοιο δικαίωμα αναβάλλεται για αργότερα ή παραμένει ακρεμές, πρέπει να δούμε ε, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων τι γίνεται με τις interim measures, με προσωρινά μέτρα πριν να είναι μια κατάσταση οριστική. Τώρα, όσον αφορά το θέμα της, ε, του εκπατρισμού, του επαναπατρισμού, της εκδίωσης, το ελάχιστο που μπορεί κανείς να συνάγει από τα αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου παρά το γεγονός ότι τα πράγματα δεν είναι πάντα πολύ σαφή διότι πολλές φορές ε, λέγεται ότι οποιαδήποτε προσφυγή ε, πρέπει να έχει ανασταλτικό ε, χαρακτήρα Πρέπει να πούμε ότι θα πρέπει κάτι τέτοιο να συμβαίνει, αλλά δεν είναι η προσφυγή η οποία θα πρέπει να έχει ανασταλτικό χαρακτήρα. Ανά πάσα στιγμή θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα όταν ζητά κανείς άσυλο να μπορεί να του εφαρμόζεται προσερινά κάποιο άλλο μέτρο θερυπίν για να μην εκδιώκεται. Δηλαδή να υπάρχει αν θέλετε, μία πρώτερη απόφαση πριν να ληφθεί η οριστική απόφαση. Μπορούμε λοιπόν να θεωρήσουμε ότι όταν μία τίθεται σε ένα αμφιβόλο μία αρνητική απόφαση για την χορήγηση προστασίας, δεν έχει αυτόματο χαρακτήρα για οποιαδήποτε προσφυγή, αλλά μπορεί κανείς να ζυγίσει, να ζητήσει, να έχει η απόφαση αυτή ανασταλτικό χαρακτήρα προσωρινά μέχρι να ληφθεί μια οριστική απόφαση. Και όταν μπορεί κανείς να δει την οδηγία, θα δει ότι παραπέμπει στο δίκαιο κάθε χώρας, το οποίο βεβαίως πρέπει να συνάδει με το διεθνές δίκαιο, με την ομολογία των δύο δικαστηρίων. Άρα δεν υπάρχει κάτι το συγκεκριμένο το οποίο να ε- το εγγυώνται όλα τα δίκαια και να είναι κοινό. Στη νέα οδηγία προτείνεται από την Επιτροπή και αυτό είναι κάτι το οποίο πιστεύουμε για ότι θα πρέπει να ισχύει για να είναι αποτελεσματική η προσφυγή σε περίπτωση ανασταλτικού χαρακτήρα, ότι θα πρέπει να υπάρχουν κάποια ελάχιστα προαπαιτούμενα για την ε, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, να θα συμφωνήσει και στις περισσότερες περιπτώσεις το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Δηλαδή, όταν έχει ε, δεν έχει ακόμη σύμφωνα με επιτυχημένη διαδικασία ε, ε εξεταστεί ένα αίτημα προσφυγής η προσφυγή θα έχει αυτομάτως ανασταλτικό χαρακτήρα. Σε άλλες περιπτώσεις, τα κράτη-μέλη μπορούν να μην προβλέψουν αυτόματα την προσφυγή, αλλά θα πρέπει να έχουν μια διαδικασία που θα του επιτρέψει να ζητήσουν τον ανασταλτικό, την αναστολή, τον ανασταλτικό χαρακτήρα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα ισχύει μέχρι να ληφθεί η απόφαση του δικαστηρίου. Τρίτη αλλαγή που προτείνει η Κομισιό, όσον αφορά τι διαδικασίε για τα σύνορα, είναι ανασταλτικές ακόμη και όταν ε, πρόκειται για υποθέσεις οι οποίες φαίνεται για όλους πρόφανες και στον κατάλογο των διεθνών προδιαγραφών ικανών, αν θέλετε, και standards, βλέπουμε ποια θέματα είναι αυτά τα θέματα τα οποία έχουν κάποια αμφισημία πολιτική, ποια θέματα είναι θέματα κάτω από τα οποία είναι κατόφλη κάτω από τα οποία δεν μπορούμε να πάμε και τι πρέπει να εφαρμοστεί. Θεωρούμε λοιπόν ότι στην πρόταση της Επιτροπής θα μπορούσαμε να συζητήσουμε ακόμη περισσότερο το θέμα αλλά δεν μπορούμε να κατέβουμε κάτω από το κατώτερο κατόφλι. Από νομικής πλευράς αυτό είναι κάτι το οποίο έτσι προβλέπεται. Τώρα, όσον αφορά την νομική συνδρομή, δίνω το λόγο στην κυρία Σαρολέα. Ήμουν αρκετά σύντομη προηγουμένως. Σας είπα ότι τίθεται δύο θέμα. Ο υποχρεωτικό χαρακτήρας από πλευρά πλευράς παροχής νομικής βοήθειας ε, δωρεάν και δεύτερον κατά πόσον αυτό είναι η καλύτερη λύση. Το πιο κατάλληλο πράγμα πρέπει να γίνει. Αυτά για τους ετούντες άσυλο. Απ' την άλλη πλευρά πρέπει να πω ότι υπάρχει νομολογία σε διάφορους τομείς που θεσπίζει δύο κριτήρια για να καθορίσει εάν ε, πρέπει να αναγνωριστεί να χορηγηθεί σε κάποιον η δωρεάν νομική αρρωγή. Ένα από τα πρώτα κριτήρια είναι, ένα τρίτο κριτήριο θα έλεγα υπάρχει. Το πρώτο κριτήριο είναι αν ο χρήστης είναι αδύναμος αν θέλετε, όσο πιο αδύναμος είναι έναντι της δικαιοσύνης, πράγμα το οποίο ισχύει κυρίως για τους ετούντες άσυλο, τόσο περισσότερο θα πρέπει να του χορηγείται η χορηγή. και δεύτερον, ποια είναι η φύση του αμφιλεγόμενου δικαίου όταν πρόκειται για κάτι το θεμελιώδες, κάτι δηλαδή το μπορεί να θέσει εν κινδύνο βασικά δικαιώματά του, ε, προστασία από βασανιστήρια, κίνδυνο της ζωής του κτλ. Ο βαθμός προστασίας, αν θέλετε, ε, θα πρέπει να είναι πιο υψηλός, αν θέλετε. Και αυτό είναι κάτι το οποίο κατά τη διάρκεια της δικαιοδοτικής διαδικασίας πρέπει να είναι σαφές. Τώρα, για θέματα ε, διοικητικά δεν είναι ίσως απόλυτα τα πράγματα σαφή. Συζητούνται όμως περαιτέρω τα πράγματα και θα πρέπει να δούμε, όχι για να είμαστε γενναιόδοροι, αλλά κατά πόσον μπορούμε να είμαστε και αποτελεσματικοί σε αυτά που κάνουμε. περισσότερε αναλύσει που έγιναν όσον αφορά τι εγγύσει τη διαδικασία για του ετούντε άσυλο σε διοικητική φάση αποδεικνύουν ότι σε διοικητικό επίπεδο, όσο καλύτερη είναι η διαδικασία, τόσο περισσότερο συμφέρει τα κράτη, διότι μειώνεται ο κίνδυνος διαπράξεως σφαλμάτων και το συστηματικό ρεφλέξε να προσφύγει κανείς τη δικαιοσύνη εάν από διοικητικής πλευράς δεν του χορηγηθεί το άσυλο το οποίο ζητά. Τώρα, το θέμα της χορήγησης ασύλου για οικονομικούς λόγους είναι διαφορετικό και βεβαίως όσο περισσότερο αποτελεσματικά μέτρα προβλέψουμε, τόσο πιο εύκολα μπορούμε να εντοπίσουμε αυτούς οι οποίοι δικαιούνται τέτοιους προστασία ή όχι. Και σε διοικητικό επίπεδο είναι σημαντικό να ακουστεί η φωνή και του ετούντος το ασύλο. Δηλαδή, στέλνει κανεί το φακελό του, αλλά είναι πολύ πιο ε, αποτελεσματικό, αν θέλετε, να υπάρχει και μια φάση συνέντευξης, να μπορεί δηλαδή προφορικά να εξηγήσει κάποια θέματα ο Τενάσιλο για να μπορέσει να ε, διαμορφώσει το αίτημά του και να σχηματίσει και πιο εύκολα εικόνα της όλης κατάστασης ε, αυτός ο οποίος καλείται να εξετάσει το φάκελό του. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε το θέμα αυτό που σας είπα όσον αφορά κυρίως τα πιο ευάλωτα άτομα που κυρίως είναι τα άτομα που ζητούν άσυλο και βεβαίως εδώ θα πρέπει να τους χορηγείται νομική συνδρομή δωρεάν. Τώρα, ε, το θέμα αυτό των ασφαλών ή σίγουρων αν θέλετε τρίτων χωρών. Θα πρέπει να δούμε κατά πόσον αυτή η έννοια είναι χρήσιμη και κατά δεύτερον να δούμε αν θα πρέπει να την εξετάσουμε από ευρωπαϊκής πλευράς η βάση εθνικών καταλόγων. Ποια είναι η χρησιμότητα αυτής της έννοιας. Απλοποιώντας κάπως, αλλά ίσως τα πιο απλά πράγματα είναι τα πιο σαφή, θα μπορεί κανείς να διαρωτηθεί. Αξίζει να διατηρηθεί μια τέτοια έννοια από τη στιγμή που θα συμφωνήσουμε με το γεγονός ότι αυτοί που ζητούν άσυλο, στους οποίους εφαρμόζεται η έννοια αυτή, θα πρέπει ούτως ή άλλως να επωφεληθούν από ένα επίπεδο διαδικαστικών εγγυήσεων σχεδόν ταυτόσιμο με όλων των άλλων πολιτών. Διότι θεωρώ πούμε ότι το ρίσκο, ο κίνδυνος, εάν ε, δεν γίνει αποδεκτή η προσφυγή, είναι θεωρω οτι το ρισκο ο κινδυνος εαν σημαντικός. Έτσι λοιπόν, θα πρέπει να δούμε πώς θα απλοποιήσουμε τις διαδικασίες. Δηλαδή, να μην χρησιμοποιούμε πάρα πολύ επαχθείς διαδικασίες για τα ευάλωτα άτομα που ζητούν άσυλο και να ζητάμε εγγύσεις δεν τις ζητάμε σε άλλες περιπτώσεις. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτή είναι η πρώτη απάντηση που μπορώ να δώσω. Δεύτερον, η ύπαρξη εθνικών καταλόγων. Μου φαίνεται ότι αυτό είναι σε αντίφαση με την ίδια την έννοια της εναρμόνισης και του ευρωπαϊκού συστήματος, δεδομένου ότι τα επιχειρήματα που αναφέρονται για να συνεχίσουν να υπάρχουν αυτοί οι κατάλογοι και κυρίως η δυνατότητα για την Ευρώπη να ενημερώνεται έγκαιρα δεν είναι πολύ πιστικό επιχείρημα από τη στιγμή που οι ευρωπαϊκές αρχές μπορούν να έχουν άμεση ε, τεκμηρίωση και να έχουν ε, τους ε, ομοιόμορφους αν θέλετε καταλόγους και κάτι που να ισχύει εξίσου με όλες, σε όλες τις χώρες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ελπίζω να μην είστε μαζί μου. Ε, δεν θα απαντήσω ακριβώς ε, μια προς μια στις ερωτήσεις σας. Θα ε, πάρει το λόγο και ο προσβήτερός μου για να απαντήσει σε όλα αυτά. Απλώς θα ήθελα να χρησιμοποιήσω το λίγο χρόνο που μας μένει για να προσπαθήσω να αναφερθώ και εγώ σε δύο ζητήματα. Το ένα το έθεσε ο εκπρόσωπος της Γερουσίας της Τσεχίας και από ό,τι κατάλαβα νομίζω ότι μιλάτε για τον μηχανισμό αναστολής του άρθρου 31 της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ρωτήσατε βάσει ποιων ε, στοιχείων θα αναστείλει τη μεταφορά προς ένα κράτος η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εάν μου επιτρέπετε, νομίζω ότι τα αίτια μπορεί να είναι, είναι μάλλον αρκετά σαφή στην πρόταση της Επιτροπής. Μιλάμε για παραβίαση διότι το επίπεδο προστασία μπορεί να είναι χαμηλότερο από τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Κάποιο μπορεί να πει ότι το εγχείρημα είναι πολύπλοκο, ότι δεν είναι ενιαίο, αλλά ιδίω γιατί τα ευρωπαϊκά πρότυπα αυτή τη στιγμή είναι, αν μπορείτε να το πω έτσι, ομιχλώδη. Όμω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να ελέγχει την ε, συμβατότητα με, τον την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία από τότε που θεσπίστηκε και από το 1977 που ιδρύθηκε δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι σε θέση να ελέγχει την συμβατότητα των εθνικών πρακτικών με τις ευρωπαϊκές διαδικασίες. Αυτό ίσως είναι μια παρατήρηση ειδικού για την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Αλλά είναι η πρώτη σκέψη που μου πέρασε από το μυαλό όταν άκουσα την ερώτησή σας. Τώρα για τις τρίτες χώρες που θα είναι την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ μία παρατήρηση. Υπάρχουν πολύ καλά παραδείγματα που αποδεικνύουν ότι μπορεί κάποιο να υποθέτει ότι ο νόμος λέει κάτι πολύ ξεκάθαρο για όλα αυτά τα περίπλοκα ζητήματα. Αλλά δεν ισχύει αυτό. Ακόμη συχνότερα έχουμε πρότυπα τα οποία επιτρέπουν κάποιες πρακτικές, σίγουρα απαγορεύουν κάποιες άλλες και μετά υπάρχουν υποσυζήτηση αμφιλεγόμενες πρακτικές βάσει των προτύπων. Η ρήτρα για τις τρίτες χώρες που είναι ασφαλείς για την Ευρωπαϊκή Ένωση από τους περισσότερους σχολιαστές θεωρήθηκε ως κατάφορη παραβίαση της αρχής για τη μη απομάκρυση, του αποπειραθώ μια απάντηση. Ή μάλλον καλύτερα να θέσω ένα ερώτημα. Η συνθήκη της Λισαβόνας τι υπενήσεται όταν λέει ότι το κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου θα πρέπει να διασφαλίζει την ε, το σεβασμό τη μη απομάκρυνση. Εννοούμε ότι το κεκτημένο το ευρωπαϊκό για το άσυλο πρέπει να διασφαλίζει ένα επίπεδο προστασία τέτοιο που να μην υπάρχουν αμφιβολίες ότι παραβιάζεται η αρχή της μη απομάκρυνσης. Διότι αν αυτό ισχύει, η ρήτρα αυτή μάλλον θα πρέπει να εξαλειφθεί από την οδηγία για τις ευρωπαϊκές διαδικασίες. Αυτός είναι ο τρόπος που αντιλαμβανόμαστε και εμείς ε, την εντολή μας. Δηλαδή, αν η συνθήκη της Λισαβόνας ορίζει ότι ο Ευρωπαϊκός Νόμος περί πρέπει να διασφαλίζει τον σεβασμό της αρχής μη απομάκρυνσης, οι αμφιλεγόμενες πρακτικές θα πρέπει να εξαλειφθούν τελείως. Και βάσει αυτού του κριτηρίου κατασκεύασα και εγώ ολόκληρη την ομιλία μου. Ίσως κάποιες πρακτικές να φαίνονται συμβατές με τα διεθνή πρότυπα, όμως υπάρχει τεράστιο περιθώριο συζήτησης όπως βλέπετε κάθε φορά. Ευχαριστώ. ευχαριστούμε πολύ με μεγάλο ενδιαφέρον αντιμετωπίζοντας το θέμα πώς αντιμετωπίζουν τα κράτη-μέλη το θέμα αυτό και τρίτων χωρών και την μελέτη για, από την ύπατη αρμοστία των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες, για τις διεργασίες που αν θυμάμαι καλά 72 χώρες είχαν εξευρεθεί και δεν υπήρχε συμφωνία ότι από τα κράτη-μέλη ότι αυτές οι χώρες ήταν ασφαλείς και μία το εν μέρη ασφαλής, μόνο όμως για άνδρες, όχι για γυναίκες και είναι και η διάσταση του φύλου που εξετάζουμε και μέσα στην οδηγία. Αυτή η μελέτη της ύπαρξης αρμοσίας ΕΕ για τους πρόσφυγες είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον σίγουρα. Κανένας νομίζω άλλος, είτε από τους εθνικούς βουλευτές είτε από τους ευρωβουλευτές δεν θέλει να παρέμβει αυτή τη στιγμή και έτσι θα κάνω κάτι το οποίο είναι ανήκουστο κάπως σε αυτό το σημείο. Θα λήξει τώρα αυτή η συνεδρίασή μας νωρίτερα, ώστε να υπάρχει περισσότερος χρόνος για ερωτήσεις, διότι ξέρω ότι θα υπάρχει ανάγκη διατύπωση ερωτήσεων υστερότερα. Λυπούμε πολύ για το ότι με αυτόν τον τρόπο θα διακόψουμε. Θέλω όμως να ευχαριστήσω όσους συμμετείχαν σε αυτό το πρώτο σκέλος και θα προχωρήσουμε μετά στο δεύτερο. Ευχαριστώ. Mesdames, Mesdames et Messieurs, Mesdames et Messieurs, nous avons gagné un peu de Κυρίε και κύριοι, έχουμε κερδίσει λίγο χρόνο. Θα σα έλεγα να συνεχίσουμε αμέσω, αφού έχουμε τέτοια ορμή. Bien, je vous propose qu'après euh, ce débat rondement mené par ma collègue Jean Lambert, nous... Μετά λοιπόν την πρωτεία Jill Lambert, ας εκμεταλλευτούμε τον χρόνο που κερδίσαμε με τη λαμπρή τη αυτή διεξαγωγή της συζήτησης για να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας αμέσως. Περνάμε στο δεύτερο μέρος λοιπόν αυτού του γύρου τραπέζης. Εγώ είμαι εισηγητής για την οδηγία σχετικά με τα ελάχιστα πρότυπα και τη δικονομία. Και περνώντα τα οριζόντια θέματα τώρα, θα έλεγα να περάσουμε σε κάποια αυτά ακριβώ τα ζητήματα που είναι πολύ άριθμα βεβαίω, αλλά θα ακούσουμε δύο παρεμβάσει αρχικά. Πρώτα απ' όλα του κυρίου Χάιλμπρονερ, καθηγητή στην, στο Πανεπιστήμιο τη ε, Κωνσταντία στην Γερμανία, ο οποίο θα μα μιλήσει για την κράτηση των, του τον άσυλο. Σας δίνω αμέσως το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, εγώ πήρα τον κλήρο να αναφερθώ ίσως στο πιο φλέγον θέμα από όλα αυτά. Η κράτηση των ετούντων άσυλο που χωρίς αμφιβολία, ακόμα και όταν όλες οι προϋποθέσεις σύμφωνα με τις προβλεπόμενες οδηγίες υλοποιούνται, είναι ένας πολύ σημαντικός περιορισμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων ενός ανθρώπου. Η νομική βάση είναι σαφής το άρθρο 5 παράγραφος 1 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Επιτρέπει μια σύλληψη ή περιορισμό ελευθερίας μεταξύ άλλων για την παρακόλληση της ε, μη, του μη επιτρεπο, εισόδου στην επικράτεια μιας χώρας. Και μετά επίσης σε σχέση με κάτι το οποίο δεν έχει εξαφανιστεί τελείως, αλλά έχουμε μια σημαντική απόφαση, την νομολογία Σάντι, όπου το ΔΕΚ, το Δικαστήριο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, ίσως προς έκπληξη κάποιων παρατηρητών, καταρχήν την παρατήρηση των Βρετανών, σύμφωνα με την οποία η σύλληψη, η κράτηση ενός ετούντος άσυλο επιτρέπεται για την αποφυγή της ε, διαφυγής του ατόμου αυτού της ε, μη επιτρεπομένης εισόδου στην ε, επικράτεια μιας χώρας. Ένα από τα κύρια θέματα που έπρεπε να απαντήσει το δικαστήριο είναι αν επιτρέπεται ένα ετών άσυλο να συλλαμβάνεται και να τίθεται υποκράτηση όταν δεν υπάρχει συγκεκριμένη επικινδυνότητα ε, συμφερόντων είτε ασφαλείας είτε άλλων δημοσίων θεμάτων ασφάλειας. Και έτσι το Δικαστήριο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Στρασβούργου έτσι, τη θέση της ε, Βουλής των Λόρδων ότι σε περίπτωση παρακόλλησης ε, ανεπίτρεπτης εισόδου και της ε, ενδυνάμει παράνομης παραμονής ενδυνάμει με, μεταναστών υπάρχει εδώ ένα ευρύ πλαίσιο διακριτικής ευχέρειας wide margin of discretion ώστε η σύλληψη, η κράτηση να μπορεί να επιτρέπεται τέτοιων ατόμων. Το σημαντικό αυτό παράθεμα θέλω να το αναφέρω αγγλικά. All that is required, όσα απαιτούνται είναι ότι η κράτηση θα πρέπει να είναι ένα αυθεντικό τμήμα αυτή της διεργασίας για να καθοριστεί αν το άτομο αυτό θα πρέπει να τύχει έγκρισης όσον αφορά την μετανάστευση ή το άσυλο. Και κατά, άλλο τρόπο δεν θα πρέπει να είναι αυθαίρετο αυτό λόγω της παραμονής, της διάρκειας, της χρονικής διάρκειας. Αυτό τι σημαίνει, ότι μόνο έλεγχος της αναλογικότητας πρέπει να γίνεται. Αν δούμε τι γίνεται στην πρακτική εφαρμογή, διαπιστώνουμε ένα τεράστιο φάσμα, τεράστιο εύρος των ρυθμίσεων για την κράτηση των ετούντων άσυλο. Υπάρχει λοιπόν ένα ευρύτατο φάσμα. Οι οδηγίες έχουν και η μέχρι σήμερα οδηγία για την διεργασία ε, χορήγησης ασύλου και της υποδοχής νομίζω πολύ σωστά καθορίζει την αρχή ότι απλά και μόνο το γεγονός ότι τίτε κάποιος άσυλο δεν επαρκεί ώστε να συλλαμβάνεται ο ετών άσυλο αν ε, δεν θα έπρεπε να κενωθεί περιεχομένου αυτή η ρήτρα, τότε η ρήτρα ότι ένα ετών άσυλο όταν δεν έχει τα αναγκαία ταξιδιωτικά έγγραφα στην ε, κατοχή του δεν μπορεί να ε, ερμηνευθεί ως επαρκής λόγος για τη σύλληψή του και την κράτησή του. Αλλά περνά τώρα στους λόγους για τους οποίους, στους οποίους προβλέπεται η σύλληψη και κράτηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε μια ολόκληρη σωρία τέτοιων λόγων. Λόγος για παράδειγμα για τον καθορισμό της ταυτότητας ή της υπηκότητας. Ο λόγος να καθοριστούν τα στοιχεία επί των οποίων βασίζεται μια ε, αίτηση ασύλου που κατά τα άλλα θα μπορούσαν να απολευθούν αυτά τα στοιχεία και η διεξαγωγή μιας διαδικασίας για την ε, έγκριση ε, χορήγησης αδείας εισόδου και η παραδοσιακή περιφρούρηση και προστασία των ε, ελευθεριών. Αυτές οι αρχές νομίζω με την ευθυγράμμιση αυτών των αρχών του ε, Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ε, του Στρασβούργου ε, είναι δεδομένη. Το θέμα είναι θα υπάρχουν περαιτέρω λόγοι, χρειάζονται περαιτέρω λόγοι. Και εδώ υπάρχει πρόταση του Συμβουλίου και θα έλεγα πραγματικά ότι θα έπρεπε να αναφερθεί, να εισαχθεί ένας λόγος ο οποίος θα αναφέρεται στο συγκεκριμένο κίνδυνο της εξαφα του να αποκριβεί το άτομο αυτό και να μην μπορεί μετά να εξευρεθεί πάλι. Absconding στα αγγλικά. Δηλαδή έχουμε εδώ τον παραδοσιακό λόγο που αναφέρεται στο άρθρο 5, εδάφιο 1, στο γράμμα F της ε, Ευρωπαϊκής Σύμβασης ε, για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, δηλαδή η ε, παρακόλληση της ανεπίτρεπτης εισόδου, αποφυγή ανεπίτρεπτης εισόδου και η αποφυγή του να εξαφανιστεί ένα τέτοιο άτομο όταν θα έχει ε, παρισφρήσει παρά, παράνομα. Και έχουμε εδώ και μια ολόκληρη σειρά διεργασιών και διαδικαστικών θεμάτων που για λόγους χρόνου δεν μπορώ να εξετάσω εδώ. Μόνο μια σύντομη παρατήρηση. Αν όλα αυτά αληθεύουν, τότε ανακύπτει ο κίνδυνος εδώ να έχουμε μια προσαρμογή, ένα συντονισμό για τους λόγους κράτησης ή ε, ε, σύλληψης μέσα στη διαδικασία κανονισμού Δουβλίνου. Έχουμε εκεί ότι επιτρέπεται η σύλληψη και η κράτηση όταν έχει ε, ληφθεί απόφαση για την μεταφορά ενός τέτοιου ατόμου. <clears throat> Κάτι τέτοιο θα ήταν περιττό αν είχαμε τον λόγο του κινδύνου του να εξαφανιστεί το άτομο αυτό. Και έχουμε εδώ το λόγο ότι μια τέτοια κράτηση επιτρέπεται όταν όλοι οι άλλοι κανόνες έχουν αποτύχει. Μου φαίνεται ότι κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό, δεν είναι ε, λειτουργικό και δεν μπορεί να είναι ε, ε, εφαρμοστέο, διότι δεν θα είναι δυνατόν πλέον να υπάρξει υπό αυτούς τους όρους κράτηση. Έτσι λοιπόν δεν νομίζω ότι κάτι τέτοιο θα ήταν μια σκόπιμη ε, διάταξη. Ένα άλλο σημείο στο οποίο θα ήθελα να αναφερθώ, ελάχιστη διάρκεια ε, μιας διαδικασίας ασύλου, ένας πολύ περίπλοκος τομέας. Δεν προβλέπεται ελάχιστη διάρκεια για την ε, εξέταση της αίτησης ασύλου. Υπάρχει φυσικά η αρχή της αναλογικότητας και δεν συμμερίζομαι τις επιφυλάξεις ε, που καμιά φορά αναφέρονται από πλευράς βιβλιογραφίας ε, ότι για παράδειγμα ο κίνδυνος υφίσταται και είναι δεδομένος τα κράτη-μέλη να καταλήγουν σε γενική, γενικά σε σύλληψη ή σε κράτηση τέτοιων ατόμων όταν δεν προβλέπεται μια ελάχιστη διάρκεια εξέτασης των αιτήσεών τους. Έχουμε διαφορετικές τέτοιες διεργασίες όσον αφορά και το δικό μας ομοσπονδιακό δικαστήριο στην ε, συνταγματικό δικαστήριο στη Γερμανία για τους λόγους για την κράτηση και πάλι εδώ έχουμε την αρχή που βλέπουμε και στο ευρωπαϊκό δίκαιο και έχει διευρυνθεί αυτό το πλαίσιο όταν υπάρχουν για παράδειγμα διοικητικές δυσχέρειες όταν επαφήνεται στην διακριτική ευχέρεια και στην ευθύνη των αρχών εδώ θα έπρεπε να δούμε αν θα είχαμε, αν θα είχαμε μια διτή ρύθμιση όπου για ένα συγκεκριμένο διάστημα, για έξι μήνες, οι λόγοι που ανέφερα θα υπαρκούσαν και μετά από αυτό το διάστημα σε ένα υψηλότερο επίπεδο θα έπρεπε να εισαχθεί μια ξεχωριστή ρήτρα κράτηση. Για παράδειγμα, λόγος για μια τέτοια κράτηση πέρα από αυτό το χρονικό διάστημα όταν υπήρξε μια απόπειρα να ε, διαφύγει ένα τέτοιο άτομο και να κρυφτεί ή όταν ε, έχουμε ε, διαδικασίες τις οποίες έχει παραβιάσει. Σύντομα δύο λόγια για την ορολογία. Δεν συμμερίζομαι τις επιφυλάξεις σύμφωνα με τις οποίες η διατύπωση δεν θα έπρεπε να καλύπτει ότι περιπτώσεις ώστε να μπορεί κανείς να καλύπτει το θέμα της μη κατανόησης της γλώσσας από τον ετούντα άσυλο, παρότι δεν είναι φυσικά η μητρική του γλώσσα αυτή. Θα έπρεπε η συμπερίληψη αυτού του όρου να θεωρηθεί ε, ότι μπορεί να συνάδει με τον κανονισμό. Στο άρθρο 9 η προτινόμενη διατύπωση όσον αφορά την πραγματική ε, νομική προστασία και όσον αφορά και την ε, κάλυψη των οικονομικών δαπανών, νομίζω ότι με την χάρτα των θεμελιωδών δικαιωμάτων συνάδει. Και μια τελευταία παρατήρηση. Όταν γίνεται λόγος ε, για πραγματική νομική προστασία και για μια χορήγηση ε, δικηγόρου ε, ώστε να μπορεί να συνδράμει ο δικηγόρος στον ετούντα άσυλο χωρίς να ε, τότε νομίζω ότι και εδώ δεν είναι το θέμα του αριθμού των ετούντων άσυλων, αλλά το 1992 είχαμε 432.000 ε, ετούντες και αν ε, με αυτού του είδους ε, την διοικητική βοήθεια καλύπτονται, τότε για όλους τους δικηγόρους θα μπορούσε να υπάρξει πεδίο δράσης, αλλά ωστόσο πρακτικό δεν είναι αυτό και δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Ευχαριστώ. Euh, Σας ευχαριστούμε. Φαντάζομαι ότι θα υπάρξουν ερωτήματα και σίγουρα και από μένα. Να δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Λοράνς Ντεμπός, η οποία είναι νομικός, ειδικό στα θέματα ασύλου και μετανάστευσης και εργάζεται στο δίκτυο Οδυσσέας και θα μας μιλήσει για το ζήτημα των ευάλωτων του άσυλων. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι. Στην παρούσα κατάφταση των πραγμάτων στο κοινότικό δίκαιο, η οδηγία για τις ελάχιστες προδιαγραφές για τους ετούντες άσυλο, που είναι η οδηγία υποδοχής, είναι το πρώτο νομικό εργαλείο πρώτης γενιάς που επιβάλλει στα κράτη-μέρη να λάβουν υπόψη την κατάσταση των ευάλωτων ετούντων άσυλο που έχουν ειδικές ανάγκες. Αυτές οι ειδικές διατάξεις, το σχετικό άρθρο σε αυτή την βασική οδηγία, επιτρέπει στα άτομα τα οποία είναι ιδιαίτερα ευπαθή και εκτεθειμένα να υποφελούνται ειδικέ συνθήκες ε, υποδοχής σε σχέση με την ειδική τους κατάσταση. Το 2007 το Ακαδημαϊκό Δίκτυο Οδυσσέας έκανε μια μελέτη για την αξιολόγηση της μεταφοράς της οδηγίας αυτής για την υποδοχή και διαπιστώσαμε ότι σε πολλά κράτη-μέλη το άρθρο 17 παρέμεινε ένα θεωρητικό άρθρο και δεν υπήρχε καμία διαδικασία ταυτοποίηση αυτών των τάπων. Ποιοι ήταν οι λόγοι. Ένας από τους λόγους ήταν ότι το άρθρο 17 αυτή τη οδηγίας στην υποδοχή δεν θεσπίζει ρητά την υποχρέωση των κρατών μελών να θέσουν σε εφαρμογή μια τέτοια διαδικασία ταυτοποίησης αυτών των ατόμων. Και αν δεν υπάρχει τέτοια διαδικασία, στις περισσότερες περιπτώσεις οι ειδικέ ανάγκες δεν μπορούν να βγουν στο φως της ημέρας, να αποκαλυφθούν. Διότι πολλοί λόγοι, αν θέλετε, δεν είναι ορατοί εκ πρώτης όψεως. Κυρίως εάν κάποιος έχει βασανιστεί, χωρίς να έχει εξωτερικά ε, στοιχεία τραυματισμού ή αν έχει υποστεί ένα κάποιο άλλο τραύμα ψυχολογικό που δεν φαίνεται εκ πρώτης όψεως. Στην νέα λοιπόν οδηγία που πηγαίνει προς τη σωστή κατεύθυνση γίνονται προσπάθειες να μπορέσει να πληρωθεί αυτή η αδυναμία, αυτό το κενό. Και αυτό είναι κάτι το οποίο χαιρετίζουμε. Το άρθρο 21 της νέας οδηγίας λέγει με σαφήνεια ότι είναι υποχρεωμένα τα κράτη-μέρη να θεσπίσουν μια τέτοια διαδικασία ταυτοποίησης, εντοπισμού. Η πρόταση της Κομισιό, παρόλα αυτά κατά την άποψή μου, θέτει ένα θέμα ενιολογικό διότι η Κομισιό δεν λαμβάνει υπόψη τον ε, ευάλωτο χαρακτήρα αυτό όπως λέγεται για κάποιες ειδικέ ανάγκες, πράγμα το οποίο μπορεί να θέσει πρόβλημα ε, σε επίπεδο νομικής ασφάλειας, αν θέλετε. Αυτό το πρόβλημα λοιπόν της έννοιας είναι ένα πρόβλημα το οποίο έγινε πιο ε, οξύ στο κείμενο του Συμβουλίου, όπου έχουμε δύο έννοιες. Ευπαθείς και ευάλωτοι ετούντες έσυλο, άσυλο και δεύτερον ετούντες έσυλο με ειδικέ ανάγκες. Και δεν υπάρχει καμία διασύνδεση μεταξύ αυτών των δύο ενιών, αν θέλετε, στο κείμενο του Συμβουλίου. Έτσι λοιπόν πιστεύω ότι το κείμενο του Συμβουλίου δεν μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη. Πρόκειται λοιπόν για ένα πρόβλημα περισσότερο τεχνικό παρά πολιτικό, το οποίο θα μπορούσε να επιληθεί σχετικά εύκολα. Εκτός από αυτό το στοιχείο, η πρόταση της Επιτροπής πιστεύω ότι θα επιτρέψει να ληφθούν περισσότερο ε, υπόψη και καλύτερα υπόψη τα προβλήματα των ευάλωτων ετούντων άσυλου ή των ετόμων με ειδικέ ανάγκες, εάν δοθούν τα απαραίτητα μέτρα για να μπορέσουν όντως οι διατάξεις αυτές να εφαρμόζονται στην πράξη. Διότι δεν είναι πάντα έτσι τα πράγματα. Έτσι λοιπόν έχουν τα πράγματα όσον αφορά το πλαίσιο υποδοχής. Τώρα, όσον αφορά την ε, ειδικέ ανάγκες των ευάλωτων ατόμων ετούντων άσυλο, όσον αφορά την διαδικασία, στην ε, οδηγία και στην ε, οδηγία του Δουβλίνου. Εδώ υπάρχει πλήρη σιωπή και οι προτάσεις κειμένου της Επιτροπής είτε πρόκειται για την ε, πρόταση οδηγίας για τη διαδικασία ή την πρόταση κανονισμού για το Δουβλίνο, τα κείμενα αυτά πρέπει να πω ότι πάνε προς την σωστή κατεύθυνση, δεδομένου ότι υπάρχουν ειδικά μέσα τα οποία ε, προβλέπονται για τα ευάλωτα άτομα ή τα άτομα με ειδικέ ανάγκες, τα ετούντα άσυλο. Το κείμενο αυτό βεβαίως ε, δεν προσφέρει τις πρακτικές λύσεις ε, όλων, για όλες τις τους ορισμούς που προβλέπονται όλες τις αρχές. Μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι η οδηγία αυτή δεν προβλέπει ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να είναι υπεύθυνα για την θέσπιση της διαδικασίας ταυτοποίησης και όπως και στην προηγούμενη περίπτωση στην οδηγία για την υποδοχή έχουμε διατάξεις οι οποίες είναι ευνοϊκές αλλά εάν δεν είναι κάτι το δεσμευτικό για να μπορέσει να τεθεί σε κίνηση η διαδικασία μπορούν να παραμείνουν ε, μόνο επί χάρτου και ευσεβείς πόθη αυτές οι ωραίες αρχές. Τώρα, αν σκεφτεί κανείς τα παιδιά αν σκεφτεί τα άτομα τα οποία έχουν ε, σοβαρά ψυχικά προβλήματα, αν σκεφτεί κανείς τα άτομα τα οποία ήταν θύματα ε, βίας, ακραίας βίας, ε, κακοποίησης, ε, βασανισμού και δούμε την διαδικασία, θα πρέπει δύο πράγματα να προσέξουμε κατά την άποψή μου είναι σημαντικά. Πρώτα απ' όλα, να δούμε ποιες είναι οι ίδιες οι διατάξεις που προβλέπει η όλη διαδικασία, διότι είναι προφανές ότι, όπως αποδεικνύουν οι διάφορες μελέτες, τέτοιου είδους τραύματα σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα συγκέντρωσης, πρόβλημα ακόμη και συμπεριφοράς κατά τη διάρκεια της συνέντευξης με το ευπαθές άτομα. Θα πρέπει αυτό να το λάβει υπόψη η όλη διαδικασία. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το λαμβάνει υπόψη η νέα οδηγία της Κομισιόν. Δεύτερον, ποια είναι η σχέση ανάμεσα στην κατάσταση ευπάθειας και τις αποδείξεις που μπορούν να υπάρχουν. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Αν δεν έχουμε την κατάλληλη διαδικασία για να μπορέσουμε να εντοπίσουμε τα διάφορα άτομα αυτά για τη διαδικασία αίτησης ασύλου, όλα αυτά τα οποία θέλουμε να κάνουμε στη θεωρία, στην πράξη θα παραμείνουν ανενεργά. Όσον αφορά τον κανονισμό του Βλήνου τώρα, το κεντρικό ερώτημα είναι το εξή. Ένα άτομα το οποίο πρέπει να μεταφερθεί κάπου, πρέπει να είναι ικανό ε, σωματικά και νοητικά να το κάνει. Μία από τις διατάξεις της ε, πρόταση τη Επιτροπή λέγει ότι μόνο τα άτομα τα οποία είναι ικανά να υποστούν αυτή τη διαδικασία μπορούν να το κάνουν. Αλλά και πάλι δεν ε, καταλήγει σε συμπεράσματα με την εφαρμογή αυτή της αρχής, διότι δεν λέγεται ποιο διαπιστώνει πότε και με ποιο τρόπο αν ένα άτομο είναι ικανό να ακολουθήσει αυτή τη διαδικασία. Τα μέσα λοιπόν δεύτερης γενιάς θέτουν το όλο θέμα αυτό για τα άτομα με ειδικέ ανάγκες που ζητούν έσυλο με εγκάρσιο τρόπο. Και αυτό νομίζω ότι είναι μια προσέγγιση που αποτελεί ένα μεγάλο βήμα προς τα μπρο. Παρ' όλα αυτά υπάρχει έλλειψη ε, ακρίβειας στα παρόντα κείμενα και έλλειψη συντονισμού μεταξύ των διαφόρων μέσων που προβλέπονται οδηγία ε, υποδοχής, οδηγία για την διαδικασία και κανονισμός του Δουβλίνου. Θα πρέπει για να μπορέσουν να εφαρμόσουν σωστά τις όλες διατάξεις και τις ειδικέ διατάξεις των τριών κειμένων να δοθούν τα κατάλληλα μέτρα στα κράτη-μέλη. Και θα πρέπει να δούμε με ποιον τρόπο θα πρέπει αυτές οι διαδικασίε εντοπισμού να εφαρμοστούν. Ε, μπορούμε να προβλέψουμε πολλά σενάρια. Μπορεί να σκεφτεί κανεί ότι θα προβλεφθεί μια διαδικασία εντοπισμού βάση μέσων και στα μέσα αυτά θα τίθενται τα ειδικά πλαίσια και μέσα σε αυτά τα πλαίσια θα καθορίζονται κάποια στοιχεία, αλλά βεβαίως μπορεί κανείς να πει ότι ένα τέτοιο σενάριο θα είναι πολύ επαχθές και δεν αποκλείει το ότι θα υπάρχουν ε, κάποιοι διάβλοι επικοινωνίες μεταξύ των διαφύρων μέσων. Ένα δεύτερο σενάριο θα είναι να κρατήσουμε το άρθρο 21 της πρότασης οδηγίας για την υποδοχή. Εγώ προσωπικά είμαι υπέρ αυτής της λύσης, διότι κατά τη διάρκεια ενός ολόκληρου χρόνου μελετήσαμε την κατάσταση σε κάποιες χώρες στις οποίες υπάρχουν τέτοιες διαδικασίες και βλέπουμε ότι πρόκειται για κάτι το πολύ ειδικό και πολλές φορές έχουμε στην πρώτη γραμμή ε, κοινωνικούς λειτουργούς, άτομα ε, τα οποία είναι τα πρώτα που έρχονται σε επαφή με αυτά τα άτομα, ενώ θα χρειαστούμε σε ορισμένε επιπτώσεις και γιατρούς, ενδεχομένως θα μπορούσαμε να έχουμε μία κοινή ε, διαδικασία και για τον κανονισμό Δουβλίνου και για τον κανονισμό διαδικασίας. Τρίτο σενάριο, να κρατήσουμε το άρθρο 21 και να σκεφτούμε ενδεχομένως ότι στην ε, ε, την υποδοχή θα προβλέψουμε έναν ενδελεχή ιατρικό έλεγχο, διότι τα περισσότερα κράτη-μέλη ούτω ή άλλω υποβάλλουν σε ιατρικό έλεγχο του ετούντε άσυλο. Αλλά εδώ θα πρέπει να είναι πιο ενδελεχή αυτό, πιο λεπτομερή αυτό ο ιατρικό έλεγχο για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις, ε, ε, στα αιτήματα των τριών ε, κειμένων εκ παραλίλου, αν θέλετε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κυρία Ντεμπός. Τελικά φτάσαμε κατά τον κανονικό μας χρόνο, πράγμα αρκετά παράδοξο. Θα δώσω το λόγο σε όσους τον ζήτησαν λοιπόν. Απρός, ήθελα να θέσω και εγώ ένα ερώτημα για τον κύριο Χάιλ Μπρόνερ και για το θέμα της γλώσσας συγκεκριμένα. Γιατί και η κυρία Ντεμπό το έθεσε σε σχέση με τα βασανιστήρια και τη δυσκολία να μιλήσει κανείς για τις περιπτώσεις βασανισμού, τι τραυματικέ εμπειρίες που έχουν ζήσει τέτοιοι άνθρωποι. Εσείς λοιπόν θα μπορούσατε να μα διευκρινίσετε τι εννοούσατε με την αναφορά σας στην γλώσσα, την γλωσσική επιλογή. Ο κύριος Ενσιού. Ευχαριστώ πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι κυρίε και κύριοι. Όταν μιλάμε για ευαίσθητε κατηγορίε του τον άσυλο, Καλό είναι να θυμίσουμε ότι υπάρχει και η περίπτωση των ασυνόδευτων ανηλίκων, των ανθρώπων με ειδικέ ανάγκε, των ηλικιωμένων, των εγγύων, των ε, ανήπανδρων γονέων με ανήλικα παιδιά, των ανθρώπων που έχουν βασανιστεί και όσο είναι θύματα σωματικής ή ψυχική βίας. Εδώ λοιπόν υποστηρίζω πλήρω την ιδέα ότι όσοι ανήκουν σε αυτή την κατηγορία του τον άσυλο θα πρέπει να είναι βασική μέρημνα των κρατών μελών γενικότερα και ειδικότερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της νομοθεσίας της. Η πράξη μας δείχνει ότι οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται από τα κράτη-μέλη στις περιπτώσεις αυτές συνήθως είναι θετικές. Δυστυχώς όμως κάποιες φορές υπάρχουν και οι είναι, είναι λιγοστές οι υποθέσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως απόδειξη θετικής εφαρμογής αυτών των διαδικασιών. Επίσης, διαφορετικές μελέτες που έχουν εκπονηθεί ως τώρα δείχνουν ότι κάποια κράτη-μέλη και επειδή ανησυχούν για μερικές μόνο από τις κατηγορίες τις οποίες ανέφερα, ιδίως για του ασυνόδευτους ανηλίκους, δεν καλύπτουν τους πάντες. Ούτε μπορούμε να μιλήσουμε το γεγονός ότι η πρόταση οδηγίας σε σχέση με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τη δικασία χορήγησης και προστασίας των Εθνικών Συστημάτων Ασύλου στα άρθρα 20 και 21 θέτει το εξή θέμα βασικό. Ιδιαίτερη προσοχή για τους ασυνόδευτους ανηλίκους. Οι υπόλοιπες κατηγορίες δεν διευκρινίζονται. Νομίζω λοιπόν ότι είναι σημαντικό το πρόβλημα αυτό να το μελετήσουμε, να λάβουμε μια κοινή θέση και να επεξεργαστούμε τα κατάλληλα κριτήρια για να μπορέσουμε να επιδιώξουμε την λύση του κάθε κάτω θα πρέπει να αναλάβει τις υποχρεώσεις του έναντι των ευάλωτων κατηγοριών του άσυλο και να αποδείξει ότι είναι αλληλέγγυο με τις χώρε ιδίω τη Ευρωπαϊκή Ένωση, βεβαίω, αλλά και αυτέ όπου το σύστημα ασύλου είναι υποπίεση. Ακόμη και αν όλα αυτά μπορούν να εφαρμοστούν μόνο σε ελούσια βάση για την ώρα και δεν μπορεί να γίνει καταναγκαστική εφαρμογή του. Σα ευχαριστώ. Θέλετε να απαντήσετε αμέσω, γιατί θα ακούσουμε ευθύ αμέσω και το επόμενο ερώτημα. Νομίζω ότι το θέμα των εξανοδευτών ανηλίκων είναι πραγματικά ευαίσθητο ζήτημα. Πολύ σοβαρό. Μπορείτε, αν θέλετε, να αντιδράσετε αμέσω και μετά το λόγο θα έχει η κυρία Ένστ κύριος βουλευτής μίλησε για έναν κατάλογο, αναφέρατε λοιπόν τον κατάλογο αυτό και η αλήθεια είναι ότι λόγω του χρόνου που μου δόθηκε δεν μπόρεσα να αναπτύξω πλήρω το θέμα αυτό, όμως ένας κατάλογος ανοιχτός, ένας κατάλογος που δεν έχει κλείσει δηλαδή. Δεν είναι κλειστός ο κατάλογος αυτός, επιτρέπει λοιπόν να καλύψουμε όλα τα άτομα, όλα τα πρόσωπα που θα μπορούσαμε να ορίσουμε ως ευάλωτα Ασχετά με το αν ανήκουν σε μια συγκεκριμένη κατηγορία, όπω τα ατομικέ ανάγκε, οι ηλικιωμένοι, ανήλικοι κ.ο.κ. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό είναι ένα πρώτο στοιχείο το οποίο καλό είναι να υπογραμμίσουμε. Σε κάθε περίπτωση και οπωσδήποτε στα πλαίσια τη οδηγία για τι ε, συνθήκε υποδοχή, για τι προποθέσει μάλλον υποδοχή, γιατί στην οδηγία για την δικονομία το ζήτημα αυτό είναι κλειστό, έχει κλείσει συζήτηση. Στην άλλη λοιπόν οδηγία αναφέρεται ιδιαίτερη προσοχή που μπορεί να αποδίδεται στους ανηλίκους, ιδίως τους ασυνόδευτους. Τόντι, τα κείμενα που χρησιμοποιούσαμε για τη μελέτη μας αποδεικνύουν ότι υπάρχει ιδιαίτερη προσοχή προς τους ανηλίκους, τους ασυνόδευτους ανηλίκους και άλλη μια κατηγορία που ανέφερα εν συντομία στην ομιλία μου, τα θύματα βασανιστήριων. Νομίζω ότι αυτό δικαιολογείται από το περισσότερο ευάλωτο χαρακτήρα. Βεβαίω είναι δύσκολο να καθορίσει κανεί ε, μια κλίμακα ευαλώτου. Όμω ένα παιδί το οποίο βρίσκεται κατάμονο και βεβαίω λόγω τη ε, ηλικία του σίγουρα βρίσκεται σε αυξημένο στάδιο ευάλωτου. ξερουμε εδω βεβαίως ότι κάποια κράτη-μέλη δεν αναγνωρίζουν τις κατηγορίες ευάλωτων ετών άσυλο. Μόνο ορισμένε. Θα συμφωνήσω λοιπόν μαζί σας. Πρόκειται για μια διαπίστωση που και εμείς ε, κάναμε στη μελέτη μας του 2007. Υπάρχουν πράγματα κάτι μέλη όπου οι ευάλωτοι δούντες άσυλο καλύπτονται και προστατεύονται λίγο πολύ ικανοποιητικά Κάναμε και μια μελέτη όπου συμμετείχαν αρκετέ χώρε. Είχαμε μια θετική αποτίμηση της στη μελέτη μα και εκεί αναφέρονται κάποιε καλέ πρακτικέ τι οποίε θα σα καλούσα να κοιτάξετε. Μερικέ είναι απλέ στην εφαρμογή του, δεν είναι αναγκαστικά δαπανηρέ και βοηθούν στον εντοπισμό των ευάλωτων ατόμων. Όμω υπάρχουν και κράτη που, πώ να το πω, ε, δεν λαμβάνουν υπόψη του όπω θα όφυλαν τι ειδικέ ανάγκε των ε, ευάλωτον ετούντων. Je change de plan <laughs> pour Ας αλλάξουμε σχέδιο. Το ρόλο έχει από την Αυστρία. Ναι, αξιότιμες κυρίες και αξιότιμοι κύριοι. Αναφέρθηκε εδώ η διαδικασία κατελάχιστον και εγώ θεωρώ ότι καλούμαστε οι διεργασίες αυτές να είναι το, οι συντομότερες ώστε γοργά να καταλήγουμε σε ένα αποτέλεσμα όσο πιο σύντομες είναι οι διεργασίες τόσο πιο ανθρώπινες είναι για τον ετούντα άσυλο για τους ανθρώπους γενικότερα γι' αυτό είναι σημαντικό για μένα οι ετούντες άσυλο να μπορούν να συνδιαμορφώνουν τη διεργασία αυτή ώστε να καταλήγει γοργά σε ένα αποτέλεσμα χειροπιαστό. Δεν βλέπω να υπάρχει κάποιο πρόβλημα, παρότι πιστεύω ότι μάλιστα είναι και πολύ σημαντικό κιόλας να καταφέρουμε εμείς τον το πεδίο παραμονής ε, ενός ετούντο άσυλο να μπορούμε να ε, το καθορίσουμε ίσως και περιοριστικά για να μπορεί να εξευρεθεί μια λύση. Δεν είναι όμως σκόπιμο να δώσουμε συνέχεια σε τέτοιου είδους σκέψεις αν θέλουμε να καταλήξουμε σε ένα ενιαίο σύστημα ε, για το άσυλο στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Να δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Ernst που το ή άλλως κάποια στιγμή θα έρθει και στο βήμα. Θα σε ευχαριστώ πολύ. Δύο ερωτήσεις, δύο θεματικά πλέγματα εδώ υπάρχουν. Το ένα αφορά την κράτηση, η σύλληψη, όπου έχω πολύ μεγάλα προβλήματα με μια τέτοια προσέγγιση και δεν είμαι και η μόνη, πιστεύω εγώ, που αυτή την προσέγγιση την θεωρεί δυσχερέστατη και προβληματική. Και είπατε κύριε Χάιλμπρόνερ, εσείς ο ίδιος, ότι θα θέλατε να είχατε και έναν πρόσθετο λόγο για παράδειγμα τον κίνδυνο να εξαφανιστεί ο ετών άσυλο. Και επισηματολογήσατε και είπατε ότι καταρχήν αυτό το μέσο της κράτησης θα μπορούσε να διευρυνθεί. Υπάρχουν αναλύσεις πόσο δαπανηρό είναι κάτι τέτοιο, για παράδειγμα στα κράτη-μέλη ερώτηση. Δεύτερον, το δεύτερο που θα με ενδιαφέρε είναι τα άτομα που έχουν ιδιαίτερες ανάγκες και πρέπει να προστατεύονται. Εδώ πρέπει πολύ πιο προσεκτικά να εξετάσουμε αυτόν τον κύκλο ατόμων. Αναφέρατε κάποιες κατηγορίες, αναφέρατε κάποιες ευάλωτες ομάδες που πρέπει ιδιαίτερα, με ιδιαίτερο τρόπο να αντιμετωπιστούν παιδιά, ε, γυναίκες, ε, γονείς που είναι μόνοι και ε, μεγαλώνουν τα παιδιά. Πώς θα έπρεπε να καθοριστεί αυτός ο κύκλος ατόμων και ποια προστασία θα έπρεπε να τους δοθεί. Περί τίνος πρόκειται συγκεκριμένα και χειροπιαστά και για ποιο λόγο αυτή η ταυτοποίηση αναφέρθηκε και απαιτείται αποσαφήνιση για αυτό τον κύκλο ατόμων. Μπορείτε ίσως με ένα παράδειγμα να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 για την ε, κράτηση Χελμπράνερ για τους λόγους. Θα έλεγα πρέπει να διαφοροποιήσουμε μεταξύ της κράτησης και του περιορισμού της ελεύθερης κυκλοφορίας. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας ότι είναι απαραίτητο να έχουμε ένα σωστό μέσο στα διάθεσή μας ώστε αν χρειαστεί να περιορίζεται το πεδίο αυτό ε, κυκλοφορίας ώστε να, για να αποφύγουμε ας το πω έτσι αφαίρεση δικαιώματος πρέπει να υπάρχει ένα μέσο ώστε να μην εντάσσεται αυτό στην κλασική αφαίρεση δικαιώματος κυκλοφορίας αλλά στο περιορισμό ε, παραμονής σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Αυτό είναι απαραίτητο ώστε να μπορέσουμε τον στόχο να τον πετύχουμε με γοργή διαδικασία σε σύντομο χρονικό διάστημα να καταλήξουμε σε διευθέτηση συζήτηση αυτών των περιπτώσεων. Φυσικά δεν είμαι ε, υπέρ του ότι θα έπρεπε να διευρυνθεί η διάσταση των λόγων ε, ε, αφαίρεσης της ελευθερίας των ετούντων άσυλο. Το αντίθετο μάλιστα κιόλας. Πιστεύω ότι θα πρέπει να περιοριστεί το εύρος αυτό των λόγων για την κράτηση. Αυτό ακούγεται ίσως ως αντίφαση. Όμως πιστεύω θα ήταν πολύ πιο σημαντικό αν καταφέρναμε να καθορίσουμε, πράγμα το οποίο θεωρώ σωστό, ότι πρέπει να υφίσταται ειδικό και ιδιαίτερο λόγο. Ότι δεν μπορεί να υπάρξει δικαιολογία ότι απλά και μόνο επειδή έθεσε κάποιος μια αίτηση ασύλου να δικαιολογείται η αφαίρεση της ελευθερίας του και να δικαιολογείται η κράτησή του. Πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι ώστε ένας ετών άσυλο να στερείται της ελευθερίας του ή να κρατείται, να συλλαμβάνεται. Ε, τότε πιστεύω να στοχεύουμε, η προσπάθειά μας να είναι να εξετάσουμε την αρχή της αναλογικότητας, να αναπτύξουμε διεργασίες και τρόπους να αξιολογήσουμε τα τα πράγματα σωστά, πρέπει να είναι serious, να υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι, να υπάρχουν συγκεκριμένοι κίνδυνοι και σοβαροί κίνδυνοι να εξαφανιστεί κάποιο ω ε, ετών άσυλο. Ε, Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί προσχηματικά ώστε συλλήβδην οι ετούντε άσυλο να ε, τίθενται υποκράτηση και να αφαιρείται η ελευθερία του. Δεν γνωρίζω αν υπάρχουν στατιστικά ή εμπειρικά κάποια στατιστικά στοιχεία για το κόστος που προκαλείται για την ε, ε, κράτηση των ετούντων άσυλο ή για την ε, στέγασή τους ή τουλάχιστον ποιο είναι το κόστος το οποίο προκαλείται από αυτές τις διεργασίες. Δεν έχω στοιχεία συνολικής ανάλυσης του κόστους που προκαλείται. Ευχαριστώ. Sur la deuxième partie la, question des catégories dans la vulnérabilité et de... Ευχαριστώ για αυτές τις κατηγορίες και για την προστασία. Κυρία Ντομπός, τι είχε να πείτε. Όντω, στο ερώτημά σα υπάρχουν δύο σκέλη. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να προσπαθήσουμε με ένα παράδειγμα πώς μπορούμε να ταυτοποιήσουμε κάποιες κατηγορίες, να τις εντοπίσουμε. Θα πάρω εγώ δύο-δύο αντίθετα παραδείγματα. Αφενός, είμαστε στην κατηγορία των ευαλώτων ατόμων τα παιδιά. Ένα μικρό παιδάκι μπορείτε να εντοπίσετε αμέσως. Απριόρι λοιπόν είναι ένα ευάλωτο άτομο. Τι είδου προστασία χρειάζεται ένα τέτοιο παιδί. Εξαρτάται αν συνοδεύεται ή όχι, ή αν είναι ασυνόδευτο. Και αν είναι ασυνόδευτο, πρέπει να βρεθεί ένας εκπρόσωπός του. Και θα πρέπει να το στεγάσουμε και να του προσφέρουμε κανονικές συνθήκες ζωής για ένα παιδάκι. Δηλαδή εκτός από το να κοιμάται να μπορεί να παίζει εντός και στο ύπεθρο, να μπορεί να πάει στο σχολείο Φερρυπίν. Να τα βασικά που χρειάζεται. Τώρα, ας πάρουμε την περίπτωση ενός ατόμου το οποίο ήταν θύμα βασανισμού. Στα πλαίσια της μελέτης που κάναμε, εδώ και ένα χρόνο συνεργαστήκαμε με 7 χώρες που έχουν προχωρήσει περισσότερο από κάποιες άλλες στα θέματα αυτό της ταυτοποίησης ή από νομοθετικής πλευράς ή στην πράξη. Και αυτό που διαπιστώσαμε είναι το εξή. Οι διαδικασίες εντοπισμού και ταυτοποίησης που λειτουργούν σωστά είναι αρκετά άτυπες αν θέλετε. Δηλαδή, περιλαμβάνουν ένα άτυπο αν θέλετε και ένα επίσημο σκέλος. Τι εννοώ άτυπο. Όταν ο, τον άσυλο είναι σε ένα κέντρο υποδοχής, έχουμε άτομα που τα περιβάλλουν, έχουμε τις κοινωνικές λειτουργούς που είναι κάπως πιο ευαισθητοποιημένα, διότι η κατάρτιση του προσωπικού και η ευαισθητοποίηση του συνόλου των, των μελών του προσωπικού είναι πολύ σημαντικό και έτσι μπορεί να δημιουργηθεί πιο εύκολα μια σχέση εμπιστοσύνης με τον ετούντα Τώρα, τα άτομα που έχουν ζήσει κάποια τραυματική εμπειρία. Ίσως κατά τη συνέντευξης ε, δεν μπορούμε να θέσουμε το ερώτημα είσαστε θύμα ε, βίας και βασανισμού ε, και δεν μπορούμε να απαιτήσουμε απάντηση. Ίσως σιγά σιγά θα μιλήσουν για τα βιώματά τους και θα αποκαλύψουν κάποια πράγματα. Βεβαίως θα πρέπει πάντα να υπάρχει διαφάνεια και από νομικής πλευράς ε, σαφήνεια απόλυτη και θα πρέπει αυτά τα δύο, το άτυπο και το τυπικό να τα συνδυάσουμε. Κάποιος ο οποίος είναι θύμα βίας ή κακοποίησης. Εάν το επιθυμούν μπορούν να τύχουν και ψυχολογικής υποστήριξης όταν πρόκειται για άτομα με ειδικέ ανάγκες ή κάποιος ανάπηρος, κάποιος που έχει χάσει που δεν έχει ε, πόδια φερρυπίν θα πρέπει να μπορεί να έχει μία αναπηρική καρέκλα ή να τον στεγάσουμε σε ισόγειο για να μην έχει να ανεβαίνει σκαλιά. Πολλές φορές κάποια πράγματα είναι αυτονόητα, κάποιες άλλες ίσως για κάποιους όχι. Θα πρέπει λοιπόν να προσπαθούμε να συνδυάσουμε όλα αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ. Η κυρία Φλότ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να επανέλθω σε ένα από τα θέματα που τέθηκε το θέμα της κράτησης. Η συνάδελφος κυρία Έστη ίσως δεν κατάλαβε στην ε, μητρική σας γλώσσα αυτό το οποίο είπατε, αλλά κι εγώ ίσως κάποια στιγμή νόμισα ότι ζητάτε συμπληρωματικά στοιχεία για να νομιμοποιηθεί αυτή η κράτηση. Πολλές φορές Καταλαβαίνετε ότι αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε πρέπει να είναι αποτρεπτικό. Το πρόβλημα το δικό μου και πολλών άλλων συναδέλφων είναι να προσπαθήσουμε να βρούμε τα κατάλληλα εργαλεία που θα μας επιτρέπουν να ελέγχουμε την χρήση από τα κράτη-μέλη τέτοιων τύπων κράτησης για άτομα τα οποία είναι ευάλωτα, που ζητούν ε, προστασία, που έχουν υπάρξει θύματα κακοποίησης και βασανισμού και δεν θέλουμε να υφίστανται ένα συμπληρωματικό βασανιστήριο αν θέλετε, να κρατούνται σε τέτοιου είδους κέντρα με συνθήκες οι οποίες δεν είναι και τόσο ανθρώπινες. Αυτό λοιπόν το διπλό έλεγχο θέλουμε να κάνουμε και αυτό σας, ε, σας ερωτώ. Ποιες είναι οι εγγύσεις οι οποίες προτείνετε εσείς να υπάρχουν για να μπορούμε να ελέγχουμε τέτοιου μηχανισμούς. Τώρα, όταν κάποιο άτομο κρατείται, ποιες είναι οι διαδικαστικές εγγύσεις ώστε να μπορεί κανείς να τους εξηγήσει σε μια γλώσσα που καταλαβαίνουν και όχι σε μια γλώσσα που ενδεχομένως θα μπορούσαν να καταλάβουν τις δυνατότητες προσφυγής που έχουν σε σχέση με την κράτησή τους και τις συνθήκες προσφυγής ή ε, χορήγησης δωρεάν διερμηνέα ή νομικής αγορογής για να μην γίνονται καταχρήσεις. Επίσης, τέθηκε το θέμα του κόστους. Πολύ σωστά. Το ε, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το θέμα αυτό του κόστους το παίρνει σοβαρά υπόψη και κάνει μία μελέτη και βλέπει και διαπιστώνει ότι τα κράτη που φωνάζουν ότι πω πω θα μας κοστίσουν πάρα πολλά χρήματα όλα αυτά προβλέπετε είναι τα κράτη-μέλη τα οποία όντως ε, για τα οποία η διαδικασία ασύλου είναι αν θέλετε πιο δαπανηρή διότι έχουν κέντρα κράτηση περισσότερο από όλου και με πολύ εύκολο τρόπο αμέσως στέλνουν σε κάποιο κέντρο κράτηση του ετούντες άσυλο. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Ευχαριστώ. Θέλετε να απαντήσετε, φαντάζομαι, για να δώσετε περαιτέρω εξηγήσει, ε, λέει η Πρόεδρο, στον κύριο Χέλμπρου. Ναι, μπορώ μόνο να επαναλάβω τα επιχειρήματά μου. Επανειλημμένα την αρχή της αναλογικότητας την τόνισα. Και είναι αυτονόητο αυστηρός έλεγχος της αρχής της αναλογικότητας απαιτείται επ' αυτού. Ίσως υπάρχει κάποια παρανόηση. Δεν θέλω να υπάρξουν οποιοδήποτε περιορισμοί ή υποβάθμιση της αρχής της αναλογικότητας. Με κανένα τρόπο. Ωστόσο αληθεύει ότι η αναλογικότητα είναι κάτι το οποίο πρέπει να εξειδικευθεί πιο χειροπιαστά. Και δύσκολο θα ήταν για μένα, το ομολογώ, ένα σετ, ένα εύρος αρχών για όλα τα 27 κράτη-μέλη να το προτείνω και ακριβώς εξειδικευμένα σημείο προς σημείο να παριθμίσω. Αλλά γιατί έχουμε ανεξάρτητα ανεξάρτητα δικαστήρια. Αυτά τα ανεξάρτητα δικαστήρια και κινούμε ότι από το ότι λειτουργούν τα δικαστήριά μας και αυτό σίγουρα θα είναι ένα θέμα για αυτά. Και ακριβώς από το, την υπηρεσία υποστήριξης ε, ε, ασύλου, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία στη Βαλέτα, στη Μάλτα, τέτοια πράγματα θα πρέπει να εξετάζονται. Στη Γερμανία δεν έχουμε υπερβολική επιβάρηση. Υπάρχουν σίγουρα προβλήματα με την σύλληψη και κράτηση ετούντων άσυλο. Αλλά δεν έχω κάποιο λόγο ή κάποια αφορμή. Ίσως ε, μπορεί να είμαι προκατηλημένος γιατί ήμουν δικαστή στο παρελθόν. Αλλά δεν έχω κάποιο λόγο να δυσπιστώ έναντι των δικαστών ότι αυτά τα μέσα τίθενται ε, σε σύγκρουση με την αρχή της αναλογικότητας ή με την αρχή του κράτους δικαίου. Για το θέμα της γλώσσας τώρα για πάλι, και πάλι είναι σίγουρα ένα επίμαχο θέμα, αμφίσιμο θέμα αν για τη γλώσσα που γνωρίζει κανείς ή αν για τη γλώσσα που εγώ έχω την, το παράθεμα στα αγγλικά ότι μπορεί να οικαστεί με εύλογο τρόπο ότι κατανοεί αυτή τη γλώσσα ο ετών άσυλο τουλάχιστον στη διατύπωση την οποία εσείς χρησιμοποιήσατε είναι μια γλώσσα κατανοητή για αυτόν. Ωστόσο θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τη διατύπωση reasonably ότι επαρκώς ευλόγως μπορεί να εικαστεί ότι κατανοεί επαρκώς ο ετών άσυλο αυτή τη γλώσσα. Λυπούμε πάρα πολύ αλλά από τη δική μου δικαστική πείρα έζησα πάρα πολλές περιπτώσεις βίωσα όπου άτομα που προφανώς κατανοούσαν επαρκώς τα αγγλικά όταν όμως εξειδικευόταν το θέμα για τους ίδιους δεν μπορούσαν να μιλήσουν ούτε μπορούσαν να παρακολουθήσουν τη διαδικασία στη γλώσσα αυτά και αυτή και αυτό δυσχέραινε τη δικαστική, διεργασία, τη δικαστική διαδικασία. Τώρα, για το αν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια γλώσσα για την οποία εύλογα μπορεί να υποθέσει κανείς ότι ο ή η αρμόδια ε, ο ή η εν λόγω ετών άσυλο ε, κατανοεί αυτή τη γλώσσα. Αν η ε, Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου προβλέπει ότι πρέπει να υπάρχουν υπάρχουν επαρκείς λόγοι για να αντικρούσει κανείς μια ε, διαταγή σύλληψης, για παράδειγμα, μια διαταγή κράτησης. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Όπως και στο προηγούμενο τμήμα της συζήτησης έχουμε τελειώσει λίγο νωρίτερα. Οπότε όποιος από εσά θέλει μπορεί να θέσει ε, πλέον ερωτήματα εφόσον θέλετε. Σε αυτήν την ομάδα ομιλητών όμως. Ο κύριος Ζεμότ δεν είναι ακριβώς ερώτημα, αντίδραση σε ερωτήσεις που ακούστηκαν από συναδέλφους για την οδηγία, την πρόταση τροποποίηση οδηγίας για την δικονομία. Έχω την εντύπωση ότι τα πάντα, όλοι νομίζουν ότι τα πάντα πρέπει να καλύπτονται από αυτή την οδηγία. Υπάρχουν αλλαγές που δικαιολογούνται από τις αποφάσεις είτε του ΔΕΚ είτε του Δικαστηρίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα και θεωρούνται αναγκαίε εκτός και δεν έχουμε κατά νου ότι και τα ίδια τα δικαστήρια, οι δικαιοδοσίε, τα δικαιωτικά όργανα δηλαδή αναγκάζονται να προσαρμοστούν στι ανάγκε τη πραγματικότητα. Το επισήμανε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχουν όμω και τροποποιήσει που επιδιώκονται για λόγου ισορροπία. Μέτρα που σκοπεύουν να καταπολεμήσουν τι δικονομικέ ε, παραβιάσει καταχρήσει. Προηγουμένω, πενιχθήκαμε το θέμα τη ενεργού συμμετοχή των ετούντων άσυλο στι διαδικασίε. Προτάσεις έχουν γίνει και από την Επιτροπή. Ζητάτε λοιπόν αυτοβούλως να προσδίδουν κάποια στοιχεία οι ετούντε άσυλο βάσει και το οδηγία για τις ελάχιστες απαιτήσει. Έτσι μπορεί να επιταχύνεται και η διαδικασία της εξέτασης της αίτηση. Ένα άλλο παράδειγμα είναι η τροποποίηση που προτείνεται σε επίπεδο των ε, αλλαγών και των ε, διαδοχικών αιτήσεων. Μετά την υποβολή μια τρίτη αίτηση μπορεί να εξεταστεί πολύ πιο ε, σύντομα το σύνολο των ε, διαδοχικών αυτών αιτήσεων και ανάλογα με την παραμονή του αιτούντα στον επικράτη του κάτω μέλους. Βλέποντας λοιπόν το σύνολο, κοιτά, βλέπ, διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μια πραγματική αναζήτηση ισορροπίας και για να υπάρχει καλύτερη προστασία που είναι δυνατή για τους αιτούντες άσυλο, αλλά για να μην υπάρχουν και κάποιε καταχρήσει που δεν θα γίνονται πλέον ανοιχτέ, έχοντα βέβαια πάντα κατά νου ότι θα πρέπει να γίνει ε, διαχωρισμό μεταξύ των όσων θα συζητηθούν πολιτικά και όσων από νομική άποψης δεν είναι αντικείμενο διαπραγματεύση. διότι ήδη προβλέπονται στην νομολογία του ΔΕΚ και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι δύσκολο λοιπόν να επικεντρωθεί κανεί σε ένα μόνο στοιχείο, εάν δεν λάβει υπόψη το σύνολο του συστήματο και το πώ τα στοιχεία αλληλεπιδρούν μεταξύ του. Ευχαριστούμε για αυτή την επιπλέον διευκρίνηση. Άλλε ερωτήσει ή παρεμβάσει τότε θα δώσω την ε, Προεδρία στη συνάδελφο για το τρίτο μέρο τη συζήτηση. C'est pas normal.

Hello. Shall we start? Okay. Uh, shall we start? Uh, a few words in Portuguese. Ξεκινήσουμε. Να πω δύο λόγια στα πορτογαλικά πρώτα. Καλό σας απόγευμα σε όλους σας. Το όνομά μου είναι Ρουί Ταβάρες. Είμαι ο συντονιστής της ομάδας της Ενωτικής Αριστεράς εδώ στην Ευρωβουλή και εισηγητής για τα θέματα ε, των προσφύγων και ιδιαίτερα για το Ταμείο Ένταξης Προσφύγων και ιδιαίτερα για το πρόγραμμα για τους πρόσφυγες. Έχουμε σε αυτή τη ε, διαδικασία τους ε, καθηγητές Ζακέ και την κυρία Γιακνοβιτσένια και χωρίς να καθυστερήσω θα δώσω τον λόγο στον καθηγητή Γαρνιέ που προέρχεται από το ε, Καθολικό Πανεπιστήμιο της ε, Λουβά και από τη Λιέγη εδώ στο ε, Βέλγιο και έχουμε σε διάφορα πανεπιστήμια ευρωπαϊκά. Έχει δώσει μαθήματα και στο Παρίσι και στη Γενέβη και στην Μπουζουμπούρα για θέματα που συσχετίζονται με τους θέματα αλλοδαπών, τον άσυλο, την ελεύθερη κυκλοφορία των ατόμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους πρόσφυγες. Και θα μας μιλήσει για το ποιος θα είναι υπεύθυνο και επομίζεται τις ευθύνες για τα θέματα ετούντων άσυλο όταν τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση ιδρούν εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρακαλώ, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κλείσατε την παρέμβασή σας αναφέροντας το θέμα που έχει τεθεί ουσιαστικά για τη σύντομη δική μου ομιλία. Το θέμα αυτό το έθεσε η δική σας Επιτροπή των Αστικών Ελευθεριών και μου μετεφέρθη αυτούσιο, δεν το διατύπωσα εγώ. Θα συγχαρώ μάλιστα εκείνον που στα πλαίσια της Επιτροπής σας διατύπωσε το ερώτημα κατά αυτόν τον τρόπο, διότι είναι πολύ ωραία η διατύπωσή του. Νομίζω ότι υπάρχουν τρεις όροι στη διατύπωση αυτή που είναι καλό να, τις, να τους αναλύσουμε. Ο όρος ευθύνη, ο όρος ποια που προηγείται και ο όρος όταν. Ποια η ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι των ατούντων άσυλο όταν οπότε, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη της δρούν εκτός της επικράτειάς τους. Θα σταθώ λοιπόν σε αυτούς τους τρεις όρους, αλλά βλέποντάς τους με την αντίστροφη σειρά. Ξεκινώντας από τον όρο «όταν». Πότε. When στα αγγλικά. Πότε η Ευρωπαϊκή Ένωση ή τα κράτη-μέλη δρούν εκτός της επικράτειάς τους. Και γιατί ξεκινώ από αυτό το τμήμα της ερώτησης, από αυτόν τον όρο. Διότι θα έλεγα ότι καταρχήν στα πλαίσια του διεθνούς δικαίου και του ευρωπαϊκού δικαίου Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε τα κράτη-μέλη δεν έχουν ευθύνη για να ασχολούνται με τους πρόσφυγες σε οποιοδήποτε σημείο του κόσμου. Θα γνωρίζετε την φράση αυτή που έχει συζητηθεί και εδώ και σε άλλες περιπτώσεις ότι δεν μπορούμε εδώ να δεχτούμε όλους τους φτωχούς του κόσμου. Αλλά θα πρέπει και εμείς κάτι να κάνουμε για αυτούς είναι η φυσική συνέχεια, το φυσικό σχόλιο. Πάντω, σε επίπεδο δικαίου δεν υπάρχει νομική υποχρέωση να ασχοληθεί κανείς με πρόσφυγες σε οποιοδήποτε σημείο του κόσμου. Ένα άλλο στοιχείο είναι η συζήτηση που λογικά θα κάνετε έτσι κι αλλιώ για την ηθική ευθύνη τη Ευρώπη. Θα συζητήσατε φαντάζομαι στο Κοινοβούλιο την ανάγκη δημιουργία κειμένων για το γραφείο που είναι υπεύθυνο για τη στήριξη των προσφύγων. Νομίζω πολλοί από εσά τονίσατε την ηθική υποχρέωση, την τεράστια ηθική υποχρέωση τη Ευρώπη έναντι των ετούντων άσυλο σε όλο τον κόσμο και το γεγονό ότι από στατιστική πλευρά η Ευρώπη υποδέχεται σχετικά λίγου ετούντε άσυλο. Όμω αυτό που ιδιαίτερα με ενδιαφέρει είναι νομική, η νομική ευθύνη ε, βάσει του δικαίου ποια είναι η ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των κρατών όταν δρούν εκτός της επικρατείας τους. Θα έλεγα ε, περιληπτικά και προστεύοντα προστεύοντας κάπως το ζήτημα ότι η Ένωση και τα κρατημέλη έχουν ευθύνη έναντι των προσφύγων που χτυπούν την πόρτα τους. Όμως όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μεταφέρουν την πόρτα τους αλλού, εκτός των συνόρων της Ένωσης. Και τοποθετούν την πόρτα αυτή στη Μεσόγειο, στη Λιβύη ή αλλού. Τότε οι πρόσφυγες πάλι χτυπούν στη δική μας την πόρτα. Αυτό θα πει ότι δεν υπάρχει νομική ευθύνη κατά την απόλυ... σε απόλυτους όρους, αλλά υπάρχει νομική ευθύνη όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση δρά εκτός της επικράτειάς της. Τότε, βάσει των γενικών κανόνων και βάσει του κοινοτικού δικαίου και του διεθνού δικαίου, υπάρχει ευθύνη. Και μάλιστα νομική. Δεν είναι απλώς ηθική αυτή η ευθύνη. Έρχομαι λοιπόν στο δεύτερο σημείο της ομιλίας μου. Την ευθύνη. Γιατί μιλάμε για αυτή την νομική ευθύνη τα κείμενα και ιδιαίτερω η συνθήκη της Λισαβόνας στο άρθρο 78 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφέρεται και αναφέρονται στο διεθνές δίκαιο και ιδιαίτερος μεταξύ άλλων στη Σύμβαση της Γενέβης και στην αρχή της μη επαναπροώθησης την οποία ήδη έχουμε αναφέρει εδώ. Ωστόσο, κατά τρόπο κυρίαρχο, η νομολογία τόσο των εθνικών δικαιοδοσιών όσο και των ευρωπαϊκών δικαιοδοτικών οργάνων. Θεωρούν ότι υπάρχει ευθύνη των κρατών ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφή στιγμή το άτομο εμπίπτει στη δικαιοδοσία, στην αρμοδιότητα μιας συγκεκριμένης δικαιοδοσίας. Δεν σημαίνει ότι κάποιος οφείλει να βρίσκεται επί της επικράτειας. Όμως, εμπίπτει στην αρμοδιότητα της δικαιοδοσίας αυτή τη στιγμή είναι σε επαφή με την αρχή ενός κράτους ή με μια αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι λοιπόν όταν η Ένωση προβλέπει διαδικασίες που προβλέπουν ότι κάπου στον κόσμο, στη Μεσόγειο ή αλλού κάποιες αρχές έρχονται σε επαφή, επικοινωνούν με τούντες άσυλο, προκύπτει ευθύνη της Ένωσης και υπάρχει ευθύνη της Ένωσης και των κρατών μελών. Ακόμη όμως δεν υπάρχει νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για το συγκεκριμένο αυτό ζήτημα του Ανατούν Άσυλο. Υπάρχει όμως νομολογία σε άλλους τομείς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και του Κοινοτικού Δικαίου για θέματα λόγου χάρη ανταγωνισμού, για να αναφέρω έναν μεταξύ των υπόλοιπων τομέων, ή για θέματα ε, κυκλοφορίας των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εκεί μπορεί να υπάρχει ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πρόσωπα τα οποία βρίσκονται εκτός της επικράτειάς της. Εάν υπάρχει βεβαίως επαφή, εάν υπάρχει συσχετισμός. Αυτό το λέει συχνά ε, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Αν υπάρχει συσχετισμός, η επαφή με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Τελευταία παρατήρηση, εάν τέτοια ευθύνη υπάρχει, ποια είναι αυτή η ευθύνη. Η πρώτη λέξη του ερωτήματός σας. Θα έλεγα λοιπόν ότι η ευθύνη αυτή, το ερώτημα της όπως έχει διατυπωθεί, μπορεί να αφορά και το περιεχόμενο και την μορφή. Δηλαδή, μιλάμε για συγκεκριμένη ευθύνη κατά την υλοποίηση της πολιτικής ασύλου εκτός της επικράτησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη μια και από την άποψη της μορφής μιλάμε για το πώς θα αναλάβει κανείς αυτή την ευθύνη στην ε, πολιτική ασύλου εκτός της επικράτησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για το πρώτο σκέλος, για το θέμα ουσίας και το τι διακρίνουμε σε αυτή την ευθύνη, νομίζω ότι έχει συνταχθεί σχετικά μια έκθεση και ήθελα να την χαιρετήσω γιατί το έργο το έργο της κυρίας Βουλέτα Μορανολάκη ήταν εξαιρετικό θα με στηρίξει στις απαντήσεις που θα δώσει αν δεν τα καταφέρω μόνος μου. Είναι εκείνη υπεύθυνη για τη σύνταξη αυτή τη έκθεση αυτή. Θα το γνωρίζετε και εδώ ότι όπως και στη δική σας περίπτωση και στα πανεπιστήμια πολύ συχνά κάποιος είναι εκείνος που παρουσιάζει τα θέματα αλλά κάποιος από πίσω του εργάζεται για αυτά. Η περίπτωση αυτή είναι η περίπτωση της κυρίας Μορενολάξ. Για συγκεκριμένους λόγους λοιπόν και αιτίες... Εδώ έχουμε να κάνουμε με τις αρχές επαναγκατάστασης προσφύγων που βρίσκονται σε άλλα κράτη, την, τα προβλήματα της τοπικής προστασίας, περιφερειακής προστασίας. Είναι πολλά τα ζητήματα που καλύπτει η έκθεση αυτή. Θα σταθώ σε ένα σημείο μόνο, στην επαφή την πόρτα, όταν λόγω χάρη γίνεται ένας έλεγχος στη Μεσόγειο. Νομίζουμε ότι εδώ θα πρέπει με μεγάλη να είμαστε πολύ σαφείς, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αποδεχτεί τον χαρακτήρα της, το, το χαρακτήρα της ανάμειξης που παρουσιάζουν οι μεταστανευτικές ροές. Στην πολιτική που σχεδιάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να ε, ελέγξει τις, μεταναστευτικέ τις μεταναστευτικές ροές, την πρόσβαση στην επικράτειά της. Ξέρετε ότι οι ροές αυτές ε, είναι συνθέτονται από άτομα πολύ διαφορετικά και μεταξύ αυτών υπάρχουν ετούντες άσυλο, υπάρχουν και πρόσφυγε. Αυτό σημαίνει ότι τα άτομα αυτά πρέπει να προστατεύονται σαν να βρίσκονταν ήδη πρώτων συνόρων μα, σαν να ήμασταν ήδη σε επαφή μαζί του. Και αυτό στα πλαίσια τη πολιτική που σχεδιάζουμε για να βγουν τα σύνορά μα πέραν τη επικρατεία μα. Εκεί λοιπόν θα πρέπει στι δράσει μα μέσω τη Frontex ή άλλων οργάνων να αναπτύξουμε μια πραγματική πολιτική ελέγχου της εισόδου που να είναι όμως και πολιτική προστασία των ατόμων αυτών που ενδεχομένως θα ζητήσουν την ε, πλήρη προστασία μας βάσει των κειμένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είτε αυτά είναι η Σύμβαση της Γενέβης είτε για την επικουρική προστασία. Και εν κατακλείδη, και αυτό είναι η τελευταία μου παρατήρηση, μίλησα και για το σκέλο τη μορφή πώ θα διοργανωθούμε στην πράξη, διότι κείμενα μπορούν να συνταχθούν. Δεν είναι ζήτημα αυτό. Αλλά η δυσκολία δεν θα είναι μόνο η επεξεργασία των κειμένων, αλλά και η υλοποίησή τους στην πράξη. Τι να κάνουμε λοιπόν, ώστε τα κείμενα αυτά, εφόσον μιλάμε για εξωτερήκευση κατά κάποιον τρόπο τη πολιτική ασύλου τη Ευρώπη. Πώ θα μπορέσουμε να διασφαλίσουμε και ένα βαθμό αποτελεσματικότητα. και πώ μέσω τη υλοποίηση θα δούμε αν μπορούμε να έχουμε πραγματική συνεργασία, πώ θα έχουμε ένα κοινό έργο μαζί και με τι τρίτε χώρε πέραν των σύνορων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ νομίζω ότι η Λισαβόνα μας δίνει την απάντηση. Θα θυμίσω το άρθρο 78 της Συνθήκης για την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο εδάφιο 2, στο τελευταίο του σημείο, στο σημείο Ζ λέγεται ακριβώ το εξή. Και παραθέτω εδώ το κείμενο, γιατί η αρχή τη παραγράφου λέει ότι ω Ευρωκοινοβούλιο μαζί με το Συμβούλιο υιοθετείτε τα μέτρα που απαιτούνται για το σύστημα, το ευρωπαϊκό σύστημα, το κοινό ευρωπαϊκό σύστημα για ζητήματα ασύλου και καταλήγει στο τελευταίο σημείο, το σημείο Ζ, για την εταιρική σχέση και τη συνεργασία μαζί με τις τρίτες χώρες ώστε να, να, να μπορούμε να διαχειριστούμε από κοινού τα μεταστατικές ροές ή τους ετούντες άσυλο ή την επικουρική βοήθεια. Άρα, η εταιρική σχέση ή η συνεργασία με τι τρίτε χώρες είναι η όρη κλειδιά. Εδώ φαίνεται ότι θα χρειαστεί να τεθεί σε εφαρμογή πραγματικά αυτή η θεωρητική ιδέα της εταιρικής σχέσης. Σχέση ισότιμης συνεργασίας ή συνεργασία, αλλά προ όφελο τη χώρα με την οποία έχουμε σκοπό να συνεργαστούμε. Δεν έχουμε σκοπό εδώ να διαμορφώσουμε όρου ε, συνεργασία υποτασσόμενου και κάποιου που θα κυβερνά τον άλλο. Αυτό που φαίνεται χρήσιμο είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση να ε, βρει ένα περιθώριο ουδέτερης συζήτησης για τις συζητήσεις της με τα τρίτα κράτη. Το πρόγραμμα της Στοκόλμης αναφέρεται σε αυτό το ουδέτερο περιθώριο συζήτησης. Αλλά δεν υπάρχει αυτό στα πλαίσια της πολιτικής ασύλου. Για σκοπούς διεθνούς συνεργασίας αστικό, στον τομέα του αστικού δικαίου. Ξέρετε ότι υπάρχουν κείμενα που επανειλημμένω έχετε συζητήσει Βρυξέλλε 1, Βρυξέλλε 2, Ρώμη 1, Ρώμη 2. Το πρόγραμμα τη Στοκχόλμη εδώ λέει το εξή. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο τόπο, ε, η Χάγη, με το Διεθνέ Δικαστήριο στη Χάγη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν θα πρέπει να ε, καταβάλει όλες τις δυνατές προσπάθειες για να προσχωρήσει και να συνυπογράψει τα κείμενα που προκύπτουν από εκεί. Μιλάμε λοιπόν για στενότερους ενδέσμους μεταξύ των κρατών μελών, για εντονότερη πολυμερή συνεργασία και με την συμβολή του ΣΥΠΑ της Αρμοστίας Λόγου Χάρη για τους πρόσφυγες και άλλους. Εκεί μπορεί πραγματικά να βρεθεί ένας τόπος για την πραγματική υλοποίηση της ε, αποτελεσματικές συνεργασίες μεταξύ των κρατών τη Ευρωπαϊκή Ένωση, των τρίτων χωρών και τη ίδια τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή είναι μια ιδέα για τι διαδικασίε, την πρακτική πλευρά του θέματος, την οποία θέλαμε να φέρουμε στην προσοχή σας. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σε ευχαριστώ πολύ για αυτή τη σαφή περιεκτική εισήγηση. Και είναι πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Διότι σε σχέση με μια τέτοια αυστηρή νομική προσέγγιση έχουμε και ηθικά συμπεράσματα και πολιτικά αλλά επίσης και χειροπιαστά πρακτικές ιδέες ώστε διαδικαστικά να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Δίνω αμέσως τον λόγο στη συνέχεια στην καθηγήτρια Γιακοβιτσένια, καθηγήτρια στη Λιθουανία, στην, στο Πανεπιστήμιο Μίκολας Ρομέρης. Ρομέρης. Ακριβώς ε, με αυτό το πνεύμα θα εξετάσει τα θέματα του δικαίου του ασύλου. Έχει εργαστεί για τους πρόσφυγες, έχει επίσης ε, ήταν ε, νομική σύμβουλος μεταξύ άλλων για διάφορους τομείς και θα μας μιλήσει στα αγγλικά για το θέμα του αν θα πρέπει να ευθυγραμμίσουμε την επικουρική επιπρόσθετη προστασία και τα θέματα διεθνούς δικαίου στις πρακτικές των κρατών μελών και να προβλέπουμε ίσα δικαιώματα για τους ε, πρόσφυγες. Έχετε τον λόγο παρακαλώ κυρία Γιακούλεβιτσένια. Αξιότιμε Πρόεδρε, αξιότιμοι Ευρωβουλευτές, ε, όπως ε, και ο συνάδελφος θα επικεντρωθώ στα ερωτήματα και θα θίξω δύο ζητήματα στη σύντομη παρέμβασή μου. Πρώτον, όταν κάνουμε λόγο για την ευθυγράμμιση των πρακτικών δικαίων στις πρακτικές των κρατών μελών, το θέμα είναι ποια είναι αυτά τα άτομα σε ποιους πρέπει να επεκτείνουμε αυτή τη διεθνή προστασία όσον αφορά την δευτερογενή προστασία των δικαιωμάτων τους. Και δεύτερον, αν αναγνωρίσουμε ότι αυτά τα άτομα πρέπει να προστατεύονται, ποια είναι η πρόσθετη αξία που δίδεται υπό το πρίσμα του ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ασχολείται με αυτό το θέμα. Όμως παρόλα αυτά το θέμα παραμένει ε, εύλογο και μέσα στο πλαίσιο του προγράμματος Στοκχόλμης. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με την σύντομη περιγραφή του προβλήματος προβλήματος. Όπως γνωρίζετε, το σημερινό φάσμα της προστασίας είναι περιορισμένο, επειδή δεν είναι όλα τα άτομα, δεν την χάνουν σε προστασίας και δεν εμπίπτουν μέσα στο ίδιο πλαίσιο ορισμών. Και αυτό δυστυχώς αντιβαίνει το στόχο της οδηγίας. Μια και ο στόχος της οδηγίας είναι να παράσχει ελάχιστους όρους και προδιαγραφές προστασίας σε εκείνους που έχουν ανάγκη προστασίας. Δεύτερον, όπως γνωρίζουμε υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των πρακτικών των κρατών μελών όταν εφαρμόζεται η αρχή αυτή τη δευτερογενούς προστασίας. Πράγμα το οποίο πάλι υπονομεύει τον εναρμονισμό της ε, στοχοθέτησης καθώς επίσης και την ε, ε, περαιτέρω ανάπτυξη του θέματος. Και θα ήθελα να πω ότι φυσικά να γνωρίζουμε στην ε, μελέτη επιπτώσεων της Επιτροπής αυτά τα προβλήματα. Να αναφέρω τώρα κάποια προβλήματα, κάποια με παραδείγματα ατόμων που βρίσκονται εκτός του φάσματος αυτού <clears throat> όσον αφορά την οδηγία. Και θα ήθελα να πω ότι όλα αυτά τα παραδείγματα τα οποία θα σας αναφέρω είτε θα βασίζονται σε διεθνείς υποχρεώσεις των κρατών μελών, είτε σε πρακτικές και εγγυήσεις που υφίστανται στα κράτη-μέλη. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα σύντομα να κάνω λόγο για τα άτομα, τα οποία θα πρέπει να προστατεύονται με την απόλυτη ε, απαγόρευση ε, επιστροφής ε, υπό το πλαίσιο προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι ένα παράδοξο για το ότι η προστασία αυτή όπως αναπτύχθηκε ιστορικά με τη βάση της απόλυτης απαγόρευσης του refoulement όταν δεν υπάρχουν εξαιρέσεις για κάποιες περιπτώσεις για τα άτομα αυτά. Και πράγματι, τι βλέπουμε από τις εξαιρέσεις που εγώ έχω συμπεριλάβει στην οδηγία βλέπουμε ότι υπάρχουν πράγματι κάποια άτομα τα οποία αποκλείονται από, τον, ε, από το καθεστώς του πρόσφυγα. Και δεν υπάρχει εδώ η εγγύηση της ε, δευτερογενούς προστασίας. Δεύτερον, μπορούμε να κάνουμε λόγο για άτομα τα οποία κατ' εξαίρεση θα πρέπει να προστατεύονται αν ας πούμε, δεν υπάρχει επαρκής προστασία σε σχέση με την ε, χώρα προέλευσής τους. Δεύτερη κατηγορία ατόμων που θα ήθελα να αναφέρω ως παράδειγμα ατόμων που βρίσκονται εκτός αυτής της ε, χορήγησης προστασίας υπό τους όρους αυτής της οδηγίας είναι τα άτομα αυτά που η οικογενειακή τους ζωή δεν διασφαλίζεται στις χώρες προέλευσής τους όπως ε, θα απαιτεί το από το άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης. Παράδειγμα, για παράδειγμα οικοί όσον αφορά το δικαίωμα της συμπληρωματικής προστασίας οικοί και συγγενείς που δεν την χάνουν της χορήγησης της προστασίας αυτής. Ή, για παράδειγμα, να αναφέρουμε επίσης την κατάσταση των παιδιών, ιδιαίτερα των ε, ασυνόδευτων παιδιών, που η προστασία τους δεν μπορεί να διασφαλιστεί στις χώρες ε, προέλευσής τους. Μια τρίτη ομάδα που θα ήθελα να αναφέρω είναι τα θύματα γενικότερης βίας και γενικότερων παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πράγματι, πολλές φορές ε, <clears throat> σε τέτοιου είδους άτομα υπάρχει η πρόβλεψη χορήγησης ε, δυνατότητας ε, προστασίας για ειδικέ τέτοιες περιπτώσεις. Στο επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε την προστασία, την προσωρινή προστασία αυτών των ατόμων όσον αφορά την κατάσταση έκδηλης παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις χώρες τους. Αυτό όμως κατ' όταν έρχονται ε, συλλογικά, όταν προσέρχονται ατομικά, αυτό δεν αναγνωρίζεται. Αυτό θέτει το θέμα της ε, συμβατότητας μεταξύ των μέσων ε, για το άσυλο και τις διαφορές που υπάρχουν όσον αφορά την αντιμετώπιση τους. Και τέλος, αλλά εξίσου σημαντικό, θα ήθελα να αναφέρω τα άτομα τα οποία παραμένουν εκτός του φάσματος του εύρους αυτής της ε, συμπληρωματικής προστασίας λόγω θεμάτων ερμηνείας ε, που τίθενται από τα κράτη-μέλη. Επιτρέψτε μου να δώσω ένα παράδειγμα για το, την εσωτερική ε, <clears throat> ένοπλη σύραξη. Αυτή διαφορετικά εφαρμόζεται και ερμηνεύεται από τα κράτη-μέλη ως εσωτερική ένοπλη σύραξη και άτομα τα οποία προέρχονται από χώρες όπου υπάρχει ε, έκδηλη ε, ένοπλη σύραξη πολλές φορές την χάνουν τέτοιας ε, σύραξης, ε, τέτοιας προστασίας, ενώ άλλα άτομα όχι. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση. Έχω δώσει κάποια λίγα από τα παραδείγματα ατόμων που παραμένουν εκτός του φάσματος της συμπληρωματικής προστασίας σε σχέση με την οδηγία. Θα ήθελα να στραφώ τώρα στο δεύτερο ζήτημα το οποίο προκύπτει. Ποια είναι η πρόσθετη αξία της διεύρυνσης ή επέκτασης της προστασίας όπως υφίσταται σήμερα σε πρόσθετες ξεχωριστές ομάδες ατόμων. Πρώτον, πρέπει να πω, ας αποκαλέσουμε ας την αποκαλέσουμε θεωρητική προσέγγιση ή θεωρητική βάση. Αν το ευρωπαϊκό κοινό ε, σύστημα για το άσυλο βασίζεται σε διεθνείς υποχρεώσεις βάσει διεθνούς δικαίου των κρατών μελών, τότε πράγματι πρέπει να διασφαλίσουμε ελάχιστες προδιαγραφές και διατάξεις για την προστασία εκείνων που χρήζουν αυτή τη προστασία. Επιπλέον, αν επεκτείνουμε το εύρος προστασίας ε, για τα παραδείγματα ατόμων που προανέφερα εγώ, αυτό φυσικά θα ευθυγραμμιζόταν και θα συνείδε με τις ε, αρχές ε, της ε, οδηγίας καθώς επίσης και θα δημιουργούσε πρόσθετη αξία, δημιουργώντας ένα ευθυγραμμισμένο πλαίσιο στην πρακτική εφαρμογή, στην χορήγηση ασύλου και προστασίας. Υπάρχουν και άλλα στοιχεία τα οποία δεν είναι λιγότερο σημαντικά. Για την κάλυψη ξεχωριστά ατόμων και το επίπεδο διαφορών που υπάρχει σήμερα μεταξύ των κρατών μελών. Αυτό θα πρέπει να ε, καλυφθεί, να πάψει να υφίσταται. Οι διαφορές μεταξύ εθνικού νομικού πλαισίου και των ε, πρακτικών. Ευθύ εξ αρχή αναγνωρίστηκε ω κάτι το οποίο έχει άμεση επίπτωση όσον αφορά την ελευθερία κυκλοφορία ε, των ανθρώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τούτου λεχθέντο, ο εναρμονισμό όλων των κατηγοριών ατόμων θα οδηγούσε στο να μπορέσει να ε, εποφεληθεί το πλαίσιο αυτό και για τα αντικειμενικά κριτήρια θα πρέπει να βασιζόμαστε στο διεθνές δίκαιο και να ανταποκρινόμαστε στις υποχρεώσεις του διεθνούς δικαίου. Υπάρχει ήδη στην πρακτική εφαρμογή η περίπτωση κάποιων κρατών που έχουν ήδη αναφερθεί σε σχέση με τον σεβασμό αυτών των ε, δικαιωμάτων των ατόμων αυτών υπό το πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και την χορήγηση πρόσθετου ε, δικαιώματος προστασίας. Τέλος, υπό πρακτική εφαρμογή η διεύρυνση αυτού του φάσματος για να καλυφθούν επιπλέον ομάδες ανθρώπων όσον αφορά την οδηγία δεν θα άλλαζε και πράγματι πάρα πολλά σε σχέση με τα όσα ισχύουν στα κράτη-μέλη στην πλειοψηφία των κρατών μελών για την προστασία αυτών των ατόμων και τα παραδείγματα που προανέφερα. Και ακόμα παραπάνω, όχι μόνο <clears throat> θα δινόταν, θα είχαν άδεια παραμονής αλλά επίσης και θα είχαν και πρόσβαση, θα ήταν ε, προσπελάσιμη η δυνατότητα εκπαίδευσης και κατάρτισης για αυτά τα άτομα. Ο εναρμονισμός λοιπόν αυτών των κατηγοριών και η κάλυψη αυτών των ατόμων μέσα από την οδηγία θα είχε επωφελή αποτελέσματα όσον αφορά την κατάστασή τους. Και τέλος θα ήθελα επίσης να αναφέρω ότι όλες οι κατηγορίες ατόμων για, τα οποία, για τις οποίες έκανα λόγο και ανέφερα κάποια παραδείγματα πιο πριν αναφέροντας ε, την επέκταση της χορήγησης προστασίας προς αυτές τις ομάδες όλες αυτές θα πρέπει σαφώς ε, να ε, καθορίζονται σε σχέση με τις, τους καθαρά ανθρωπιστικούς λόγους. Διότι εδώ υπάρχει και η ε, καταδιάκριση, η καταδιακριτική ευχέρεια προστασία των ατόμων αυτών που δεν καλύπτονται από τις ε, ε, διαφορετικές διατάξεις. Υπάρχουν και θέματα ατόμων που είναι υπερήλικα ή ότι όταν υπάρχουν προβλήματα όσον αφορά την απέλαση ή επιστροφή τους στις περιπτώσεις αυτές δεν ήταν αυτές που ήθελα εγώ να αναφέρω αλλά με βάση τον εναρμονισμό των διεθνών υποχρεώσεων του διεθνούς δικαίου από πλευρά των κρατών μελών καθώς επίσης και των πρακτικών που ήδη φύστανται στα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ κυρία καθηγήτρια Γιακούλεβιτσένε για την παρέμβασή σας που ήταν πάρα πολύ ενημερωτική και για το επιχείρημα το οποίο δομήσατε και παρουσιάσατε περιεκτικά και με πλήρη τρόπο και εξειδικευμένα υπέρ του εναρμονισμού της ε, συμπληρωματικής επιπρόσθετης προστασίας για αυτές τις περιπτώσεις ατόμων που είτε βρίσκονται εκτός ε, νομικού πλαισίου είτε ε, εκτός κάλυψης. Έχουμε κάποιες ερωτήσεις. Θα δώσω αμέσως τον λόγο στην συνάδελφό μου Ελέν Φλότρο από την ομάδα των Πρασίνων. Παρακαλώ Ελέν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να καλέσω τον κύριο Καρλίε να διευκρινίσει την ευθύνη που εμπίπτει στα κράτη-μέλη ή της Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια των δράσεων της Frontex που έχουν κάποιες επιπτώσεις. Παίρνω ως παράδειγμα την Λαμπεντούζα, το νησί αυτό στο οποίο υπήρχαν εκατοντάδες πρόσφυγες και μας έλεγε ο για τους πρόσφυγες ότι πολλοί θα μπορούσαν να τύχουν διεθνούς προστασίες ενώ σήμερα φτάνουν κάποιες εκατοντάδες άτομα στην Λαπεντούζα και θα ήθελα αυτή η δυνητικά ή νόμιμα ε, άσυλο που πηγαίνουν. Και εδώ τίθεται το θέμα της Frontex και των ευθυνών της. Όταν διηγούμε αυτά στον ε, ε διευθυντή Frontex δεν ανησυχεί καθόλου διότι αυτός ασχολείται με θέματα επιμελητίας και η ευθύνη είναι απλώς θέμα ευθύνης των κρατών μελών. Είναι λοιπόν σαφές ότι βεβαίως όταν αργούμε στην επικράτεια με σχόραση στα χωρικά της Ήδακα ξέρουμε τι συμβαίνει, αλλά όταν η Frontex ενεργεί εκτός χωρικών υδάτων είναι πολύπλοκο το θέμα της ευθύνης και πολύ πολύπλοκο. Γι' αυτό παρακαλώ στα πλαίσια τέτοιου είδους επιχειρήσεων, πείτε μου σε ποιον εμπίπτει η ευθύνει το θέμα της ε, ε, εφαρμογής της αρχής της επαναπροώθησης και βεβαίως είναι δεσμευτικό αυτό το οποίο λέγει ο Ευρωπαϊκός Χάρτης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, είναι δεσμευτικά αυτά που λέγονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και με την αλλαγή της όλης κατάστασης με την θέση σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας, ε, οι δράσεις της Frontex πολλές φορές είναι κάτι που μπορούμε να ελέγξουμε, αλλά σε άλλες περιπτώσεις δεν μπορούμε. Θα ήθελα λοιπόν για αυτή την κάπως ασαφή κατάσταση, με ε, επιπτώσεις όμως πολύ συγκεκριμένες για το δικαίωμα ασύλου στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια, να μου δώσετε κάποιες διευκρινήσεις. Πιστεύω ότι ε, δεν χρειάζεται να χωρίσουμε τις ερωτήσεις ε, ε, για ερωτήσεις μεταξύ ευρωβουλευτών ή εθνικών βουλευτών. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ανά δύο ερωτήσεις θα ήθελα να απαντώνται. Η Τζιν Λάμπερτ. Ευχαριστώ. Μιλήσατε για σχέσεις με τρεις χώρες. Για αυτή την έννοια της, ε, των ε, ίσων, ισονόμων εταίρων. Εμείς αυτό το θέμα δεν το βλέπουμε να είναι θέμα ισότητας ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Κάποιες χώρες ε, θέλουν να επιτύχουν συμφωνία με τη Λιβύη, Φερρυπίν, για να δώσω ένα παράδειγμα διότι πολλές φορές θεωρείται χώρα διαμετακόμιση Λιβύη, θέλουν κάποια άτομα να επαναπροωθούνται εκεί. Υπάρχουν θέματα τα οποία για μας είναι πολύ σημαντικά για να δούμε η ιατρική σχέση τι ακριβώς σημαίνει σε τέτοιους περιπτώσεις, διότι υπάρχουν και επιπτώσεις ε, και είναι και θέμα ηθικής ευθύνη και των δράσεων που μπορούμε να αναλάβουμε μετά στα πλαίσια της συνεργασίας με άλλες χώρες που βρίσκονται αν θέλετε στα σύνορά μας. Και θέλουμε να δούμε η ποιότητα της προστασίας πώς είναι. Πού βρίσκεται. Επίσης, τώρα το θέμα του, της αρχής επικουρικότητας και του καθεστώτες του ετούντος ασύλου. Ξέρουμε ότι πολλές φορές γίνεται προσπάθεια από κράτη-μέλη αυτά τα δύο θέματα να ε, ε, επιλύονται με την ίδια προσέγγιση ενώ το θέμα των ε, ελαχίστων ε, απαιτήσεων και τις, ε, στις οδηγίες των ελαχίστων απαιτήσεων είναι διαφορετικό. Εμείς είπαμε εδώ και χρόνια του Κοινοβούλιο ότι η επικουρική προστασία θα πρέπει να είναι βραχυπρόθεσμη. Είναι πραγματικότητα αυτό στις έρευνες που κάνατε, πώς το και το θέμα αυτό. Και τελικά, τι πιστεύετε ότι θα πρέπει να συμβαίνει σε άτομα τα οποία δεν είναι δικαιούχοι ανθρωπιστικής ε, βοήθεια στα πλαίσια της οδηγίας των ελαχίστων απαιτήσεων αλλά όπω λένε και κάποια κράτη-μέλη δεν μπορούν να επιστρέψουν στη χώρα προεβολή τους. Στη Ζιμπάουε, Φερρυπίνο, που υπάρχει γενικότερο κλίμα βία. Ε, και πολλές φορές έχουμε αντινομία μεταξύ εθνικού δικαίου και δικαιώματος ασύλου. Έχετε παραδείγματα τέτοιου τόπου. Πώς τα κράτη-μέλη πρέπει να αντιμετωπίσουν την κατάσταση των ατόμων που δεν ε, είναι δικαιούχοι τέτοιου είδους προτεσίες αλλά παρόλα αυτά δεν μπορούν και να επιστρέψουν στις χώρες τους. Θα ήθελα να δώσω πρώτα το λόγο στον κύριο Καρλία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρο. Σε σχέση με το θέμα της κυρίας Φλότρου. Ποια ευθύνη και μετά να δούμε πιο συγκεκριμένα τι γίνεται με τη Frontex. Σε σχέση με τον έλεγχο των ατόμων πέραν των συνόρων της Μεσογείου Φερρυπή, θα πρέπει να αναφερθούσουμε σε μια σημαντική νομολογία που ισχύει για παρεμφερείς καταστάσεις της ΕΠΑ κατάσταση των Αιτινών boat people που ήθελαν να φτάσουν στις ε, Αμερικανικές ακτές μετά από αποφάσεις που είχαν λάβει διάφορες αποφάσεις ε, ε, αμερικάνικες και οι ακτοφυλακοί οι αμερικάνικοι έλεγξαν τα άτομα αυτά πέραν των χωρικών υδάτων των ΙΠΑ. Και το κύριο επιχείρημα των ΙΠΑ ήταν ότι όταν ο έλεγχος γίνεται εκτός της εδαφικής μας επικράτειας ή εκτός χωρικών μας υδάτων δεν, είναι, δεν είμαστε υπεύθυνοι και δεν είμαστε υποχρεωμένοι να τηρήσουμε την αρχή της μη επαναπροώθησης έτσι όπως αναφέρεται στο άρθρο 32 της Σύνδεσης Γενέβης. Θα πρέπει όμως να διευκρινίσουμε το εξής. Το νότο δικαστήριο τον είπα γι' αυτό το θέμα δικαίωσε την κυβέρνηση των ΗΠΑ. Διότι είπε ότι δεν χρειάζεται να τηρήσουν την αρχή της μη επανυπρόθεσης, είπα, πέραν της επικράτειάς τους. Και θα ήθελα να πω ότι σε διεθνές δίκαιο, καθώς και είπατε αρμοστία, στο διεθνέ δίκαιο, καθώ και είπατε αρμοστία των εθνών που παρενέβησαν σε αυτή τη διαδικασία, στο σύνολό του όλοι σχεδόν κατέληξα στο συμπέρασμα ότι δεν ήταν σωστή η ερμηνεία αυτή για την μη επαναπρόθεση. Αλλά πρέπει να σας πω ότι γίναν συζητήσει και σε επίπεδο ανώτατο δικαστήριο, ότι το ανώτατο δικαστήριο τον είπα, δεν είναι οποιοδήποτε δικαιοδοτικό όργανο. Υπάρχουν κάποια θέματα εσωτερική δικαιοπαρεμβάνω, αλλά εν πάση περιπτώσει για μας τώρα, για τον Οδυσσέα, για το δικό μας δίκτυο, μπορώ να πω ότι σχεδόν ομόφωνα θεωρούμε ότι αυτή η απόφαση του Ανώτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ δεν είναι σωστή τήρηση της αρχής και σεβασμός της αρχής επαναπρόθεσης. Και αργότερα χρονικά η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΝΟΥ στα πλαίσια της ε, εφαρμογής της Διεθνούς Σύμβασης για κάποια άλλη υπόθεση θεώρησε ότι υπήρχε καταστρατήγηση της αρχής της μη επαναπρόθεσης. Και βεβαίω, ξέρουμε ότι γίνονται σε ε, νομικό επίπεδο πολλές συζητήσεις, ξέρουμε ότι υπάρχουν ε, κάποια θέματα τα οποία με απόλυτη σαφήνεια επιτρέπει ο νόμος, ε, απαγορεύει ο νόμος, αλλά υπάρχουν και κάποιες φεζόνες. Και εδώ βεβαίως θα πρέπει να τηρήσουμε οπωσδήποτε την αρχή της μη επαναπρόθεσης και πέραν των ε, εθνικής Τώρα, για τη Frontex τι γίνεται σε περίπτωση καταστρατήγης αυτού του, αυτής της αρχής από τη Frontec. Πρώτα απ' όλα, θα πρέπει να γνωρίζει κανείς πολύ καλά την κατάσταση. Γιατί το απέδειξε αυτό η, η ερώτησή σας. Σήμερα βασιζόμαστε σε εκτιμήσεις. Διότι κάποια στιγμή λέμε ότι πήγανε άπειρα άτομα στη Λαμπεντούζα Φερρυπίν, την επομένη είχαμε λίγες δεκάδες, που πήγαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Κάποια στιγμή κάνουμε λοιπόν εκτιμήσεις και βλέπουμε ότι πραγματικά χρειάζεται να έχουμε ένα πάρα πολύ καλό εργαλείο αξιολόγησης των δράσεων της Frontex σε σχέση με την αρχή της μη επαναπρόθεσης και σε σχέση με την δυνατότητα που έχουν οι ετούντες ατσιλό να ζητήσουν να τους χορηγηθεί αυτή η ιδιότητα. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει εφ' εξής, και αυτό είναι κάτι το οποίο εσείς θα πρέπει να απαιτήσετε, εφ' εξής θα πρέπει οι εκθέσεις της Frontex να περιέχουν σαφή αξιολόγηση ε, των ε, συμβάντων όταν έχουμε τέτοιου είδους ε, περιπτώσεις. Πράγμα το οποίο δεν βρίσκουμε σήμερα στις εκθέσεις που μας αποστέλει Frontex. Το ίδιο και συμβαίνει και εδώ φτάνω τώρα στην δεύτερη ερώτηση της κυρίας Λομπέρ όσον αφορά τις συμφωνίες που θα μπορούσαν ενδεχομένω να υπογραφούν μεταξύ Frontex και τρίτων χωρών. Και λέει η κυρία Λόμπερ και υπογραμμίζει το θέμα της εταιρική σχέσης που βεβαίως ε, δεν έχει ε, ε σε αυτή την περίπτωση να κάνουμε πάντα με ισότιμους εταίρους όσον αφορά την πρόσπιση κάποιων δικαιωμάτων ή την προστασία. Γι' αυτό το λόγο Πιστεύω ότι είναι αρκετά δύσκολο να πούμε εκ των προτέρων ότι μπορούμε να προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία με την χ χώρα και όχι με την ψ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πιστεύω ότι ε, η ίδια αποφασίζει ανεξάρτητα ποιε είναι οι χώρε με τι οποίε θα συνάψει συμφωνία, αλλά θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτική όσον αφορά το γενικότερο πλαίσιο ή την τήρηση των ανθρωπίνων και σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα αυτή. Όταν όμω δεν έχουμε κάτι το, όταν έχουμε κάτι το οποίο βγαίνει εκτός της απευθείας σχέσης Ευρωπαϊκής Ένωσης κρατών μελών και τρίτης χώρας μπορούμε να έχουμε από νομικής πλευράς κάποιο είδους ερωτηματικά και ανησυχίες. Εγώ βεβαίως πρέπει να σας πω ότι δεν αναφέρομαι σε θέματα διεθνούς ιδιωτικού δικαίου ή προγράμματος Χάγης. Η εμπειρία σε θέματα διαπραγμάτευσης διεθνών συμβάσεων με κάνουν να πω ότι όλες οι προπαρασκευαστικές εργασίες καταλήγουν σε συμφωνίες οι οποίες κυρώνονται σε πολύ μεγάλο βαθμό. Σκέφτομαι το θέμα της ε, σύμβασης της Χάγης για την ε, υιοθεσία παιδιών, όπου επιτρέπεται να υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ της, των διοικητικών οργάνων όχι της χώρας προέλευσης του, του πρόσφυγα αλλά της χώρας από την οποία περνάει και της χώρας η οποία υποδέχεται ε, τους μετανάστες. Μια τέτοιου είδου συνεργασία θα μπορούσε να καταλήξει καλά αποτελέσματα. Και βεβαίως θα πρέπει πράγματι να μπορεί κανείς να είναι σίγουρος ότι οποιαδήποτε διαπραγμάτευση αρχίζει μεταξύ εταίρων που είναι ε, βάσει κάποιων κριτηρίων στο ίδιο επίπεδο. Διαφορετικά μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να θέσει κάποια θέματα. Η κυρία Λακουβιτσένια. Σας ευχαριστώ πολύ για το θέμα του αν πρέπει να υπάρχουν ε, ε, ξεχωριστές ε, γραμμές ε, και κατηγορίες για πρόσθετη προστασία. Ο λόγος για τον οποίο δεν ανέφερα αυτό το στοιχείο στην παρουσίασή μου δεν ήταν μόνο λόγο του χρόνου που πίεσε. Ο λόγος είναι ότι φυσικά εμείς εκτιμούμε πλήρως αυτό που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην διατύπωση της πρότασής της Εξετάζοντα τα επιχειρήματα τώρα, φυσικά αφενό υπήρχαν κάποια επιχειρήματα κατά της, ε, ε, των διαχωριστικών αυτών γραμμών ή της εξίσωσης. Και ένα από τα στοιχεία που αναφέρατε ότι η επικουρική προστασία, η πρόσταστη η προσταστη προστασια θα παρέχεται για πολύ συντομότερο χρονικό διάστημα από ότι ε, το καθεστώς για παράδειγμα πρόσφυγα. Το άλλο επιχείρημα είναι το ότι πράγματι το άρθρο 78 παράγραφος 2 της συνθήκης για την, της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάνει μια διαφοροποίηση πράγματι μεταξύ των δύο καθεστώτων αυτών και ειδικά ιδιαίτερα για την έννοια του ασύλου το καθεστώς πρόσφυγα είναι ισχυρό πανευρωπαϊκά ενώ εδώ δεν αναφέρεται το θέμα της επικουρικής ε, ε, παροχής προστασίας. Το άλλο επιχείρημα που θα ήθελα να αναφέρω και εδώ πρέπει να πω ότι στη μελέτη μας δεν είχαμε κάποιες ε, νέες ε, αξιολογήσεις στοιχείων. Βασιστήκαμε σε μελέτες ε, στοιχείων όπως της είπα της Αρμοστίας των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες και εδώ το επιχείρημα για την σύντομη ε, διάρκεια προστασίας, ε, επικουρικής προστασίας δεν αντανακλά την ίδια την ε, πραγματικότητα, διότι αυτοί, αυτά τα άτομα μπορεί να παραμείνουν και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε μια χώρα. Το θέμα είναι το θέμα της ικανότητας αφομοίωσης ή ολοκλή... ένταξης αυτών των ατόμων σε αυτές τις κοινωνίες. Δεν μπορούν να παραμείνουν χωρίς δικαιώματα. Και έχουμε και το ότι η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην αξιολόγηση μελέτης αναφέρεται σε δύο περιπτώσεις ε, ε, από την νομολογία του ε, Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Στασβούργου όπου λέγεται ότι δεν πρέπει να υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ ατόμων που θα έχουν πρόσβαση στα επιδόματα ε, τέκνων ε, και την υποστήριξη ε, για τα παιδιά τους και έτσι να μην παραμείνουν χωρίς αυτά. Δεν πρέπει να υπάρχει διαφοροποίηση λοιπόν μεταξύ αυτών των ατόμων και άλλων που έχουν το καθεστώς μόνιμης άδειας παραμονής στην επικράτεια μιας χώρας. Και εδώ φυσικά υπάρχουν επιχειρήματα τα οποία θέτουν το θέμα ότι ενώ προσπαθούμε να πετύχουμε ένα ενιαίο καθεστώς θα πρέπει να γίνεται λόγος για ίσα δικαιώματα, ίσες και ε, ευκαιρίες σε ένα ισότιμο πλαίσιο. Και τώρα η πρακτική των κρατών μελών, δηλαδή πώς τα κράτη-μέλη αντιμετωπίζουν αυτά τα άτομα της επικουρικής ή επιπρόσθετης προστασίας ε, και σε σχέση με τα άτομα που έχουν το καθεστώς πρόσφυγα. Το μόνο το οποίο μπορώ να πω είναι, μια και δεν είμαστε εμείς εκείνοι που κάναμε αυτές, αυτά τα ερωτηματολόγια και τις συνεντεύξεις στα κράτη-μέλη, αλλά βασιστήκαμε σε αυτές τις μελέτες, είναι σαφέστατο ότι υπάρχουν διαφορές μεταξύ των κρατών μελών. Σε κάποια κράτη-μέλη μπορείτε να βρείτε σχεδόν ίσα, ισότιμα δικαιώματα μεταξύ προσφύγων και δικαιούχων επιπρόσθετης ή επικουρικής προστασίας. Σε κάποια άλλα κράτη-μέλη μπορείτε να βρείτε αναντιστοιχεία αυτών των δικαιωμάτων και αν θυμάμαι καλά και αν επιτρέπετε πρόεδρε υπάρχουν μόνο λίγα κράτη-μέλη που πράγματι καταφεύγουν καταλήγουν σε αυτές τις κατεξαίρεσιν διατάξεις ε, που επιτρέπει το σημερινό κείμενο της οδηγίας δεν υπάρχει λοιπόν ε, ε, μια ευρύτερη πρακτική, α το πω έτσι, τη επικουρική χορήγηση προστασία. Και τέλο, τι συμβαίνει με τα άτομα τα οποία δεν είναι δικαιούχα ε, επιπρόσθετη επικουρική προστασία μέσα στο πλαίσιο αυτή τη οδηγία. Και πάλι εδώ, είναι σαφές το γεγονός ότι υπάρχουν πολύ διαφορετικές πρακτικές από τα κράτη-μέλη εναντί αυτών των ατόμων. Αν κάποια κράτη-μέλη χορηγούν κάποιου είδους ανθρωπιστική, ε, ανθρωπιστική ή άλλου είδους υποστήριξη εκτός ε, της, ε, του ορισμού της επικουρικής προστασίας, κάποια από αυτά χορηγούν αυτή την υποστήριξη και μέσα ίσως και σε ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν κάποια κράτη-μέλη που καταλήγουν σε ένα αποδεκτό καθεστώς ή ανεκτό καθεστώς για αυτά τα άτομα χωρίς να τους χορηγούν ένα σταθερό καθεστώς έναντι ε, εκείνων που έχουν για παράδειγμα άδεια παραμονή στη χώρα. Υπάρχουν και κάποιες ε, πρακτικές όπου ακόμα και για αυτές τις άδειες άτομα που αποκλείονται από το καθεστώς του ε, πρόσφυγα που όμως υπάρχει εδώ η απολυτότητα του νογεφουλμό υπό τους όρους του ε, ανθρωπιστικού δικαίου των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Σε σχέση με αυτή την οδηγία λοιπόν, ας το πω έτσι, προβλέπεται ένα μεγαλύτερο πλαίσιο από αυτό το οποίο χορηγούν τα κράτη-μέλη εναντί αυτών των ατόμων. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ. Ομολογώ ότι τώρα ανησυχώ πλέον με το χρόνο. Πιέζει ο χρόνο. Έχουμε τέσσερι που ζητούν να παρέμβουν. Περνούμε αμέσω στον καθηγητή κύριο Φιλίπ Ντεμπρουκέρ. Θα είναι αδύνατο να καλύψουμε όλε τι ανάγκε μέσα στο χρονικό πλαίσιο. Αλλά δεν θέλω να υπάρξει περικοπή του χρόνου τη επόμενη ε, ε, συνέντευξη. Παρακαλώ. Δεν θέλετε να παρέμβετε. Η κυρία καθηγήτρια Λοράνς Ντεμπός, παρακαλώ. Ε, ε, Όχι. Ε, τότε από την Εθνική Συνέλευση της Σλοβενίας ο κύριος Ρόζε εδώ έχουμε ούτε κι εσείς ο κύριος Κάι Χάιλμπρον παρακαλώ έχετε τον λόγο κύριε Χάιλμπρον Um, could you please state your name because... Πείτε uh, μας το όνομά σας παρακαλώ γιατί δεν το έχω. Βιολέτα Μορένο Λάξ. Βιολέτα Μορένο Λάξ. Και σε σχέση με τον κύριο Καρλιέ είχα ε, συνεισήγηση και ήθελα να αναφέρω σε σχέση με το ερώτημα το οποίο τέθη για τη Frontex να πω το εξής για την ευθύνη της ε, Frontex θεωρητικά σε σχέση με ε, την θέση για την Frontex είναι σαφής ε, ως σώμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται η Frontex κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης ε, της εντολής της να τηρεί και να παρατηρεί και να τηρεί την, τα, τις ε, διατάξεις ε, για τη διαφύλαξη και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και μετά στην διατύπωση σε σχέση με το άρθρο 1 αναφέρεται η υποχρέωση της Frontex να ε, συνάδουν οι δράσεις της με τα θεμελιώδη δικαιώματα. Το ίδιο επίσης σε σχέση με το πρώτο τμήμα. Το πρόβλημα δεν είναι λοιπόν σε σχέση με την απαρίθμηση των υποχρεώσεων της Frontex σε σχέση με τα δικαιώματα του ανθρώπου. Το θέμα είναι το θέμα των ρητρών ασφάλειας. Αυτή αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν ε, ρήτρε ασφάλεια. Αν κάποιο ε, πρόσφυγα ή κάποιο ετών άσυλο ε, παραπονείται για τον non-refoulement, δεν υπάρχει τρόπο να υπάρξει θεραπεία για το αίτημα ή το ζήτημα αυτό, ώστε να αποκατασταθεί οποιαδήποτε ζημία υφίσταται καθιονδήποτε τρόπο θα είναι ε, θέμα το οποίο θα τίθεται αυτό όσον αφορά την ε, διατύπωση της ε, εντολής για την Frontex. Από την άλλη πλευρά για το μηχανισμό για την Λαμπεντούζα με τις, όταν αναφέρεται ότι είχαμε χιλιάδες αφήξεις στο παρελθόν και τώρα έχουμε κάποιους εκατον, κάποιες εκατοντάδες από αυτούς που πήγαν όλοι αυτοί. Έχουμε και την διαπραγμάτευση σε σχέση με τον, τον κανονισμό ΕΑΣΟ και αλλαγές που έχουν εισαχθεί και ίσως εδώ και μια ρήτρα σε σχέση με την υποχρεωτική συμμετοχή της, ε, του, της υπηρεσίας υποστήριξης για το άσυλο, Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο όσον αφορά τα θέματα αυτών των ανθρώπων. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ κυρία ε, καθηγήτρια Μορένο Λάξα. Με αυτές τις αποσαφηνήσεις λοιπόν καταφέραμε να τηρήσουμε τον χρόνο και περνάμε λοιπόν και δίνουμε τώρα στον κύριο Σάιμον Μπουσούτιλ την πρωτοκαθεδρία. Παρακαλώ για τον επόμενο γύρο. Ε, λοιπόν, εντάξει αγαπητοί φίλοι, συνεχίζουμε τις εργασίες μας με το τέταρτο τμήμα και τελικό τελευταίο τμήμα αυτής της συνεδρίασης. Έναν ομιλητή έχουμε, που είναι ο καθηγητής Henri Λαμπάιλ, καθηγητής <clears throat> στο Πανεπιστήμιο της Μπαϊόν, ε, Πανεπιστήμιο του ΠΟ μια σύντομη εισαγωγή. Είναι καθηγητής ε, δικαίου, έχει την έδρα Ζόμονε στο Πανεπιστήμιο του ΠΟ και είναι ο πρίτανης ε, της ε, ε, σχολής, της νομικής σχολής του Πανεπιστημίου της Μπαγιών. Έχει ασχοληθεί με την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, το δημόσιο δίκαιο της ελευθερίας και την κοινωνική Ευρώπη. Ο καθηγητής Λαμπάιλ θα μας αναφέρει ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Πώς το κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου μπορεί να είναι συνεκτικό και σε σχέση και με την σύμβαση της Γενέβης να, ενισχυθεί, να ενισχυθούν οι εξουσίες της υπηρεσίας υποστήριξης ασύλου ή να δημιουργηθεί και ένα δικαστήριο για θέματα ασύλου ευρωπαϊκού χαρακτήρα. Είμαι σίγουρος ότι αυτά τα θέματα θα τύχουν ορθής παρουσίας σας από τον καθηγητή Λαμπάη. Έχετε τον λόγο παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, όπως και ο κύριος Μπρινέρ. Ε, ε, επελέγει ως αυτός ο οποίος δεν θα τηρήσει το χρόνο. Πρώτα απ' όλα δεν έχω τέτοιους περιορισμούς διότι ο χρόνος έχει περάσει ούτως ή άλλως και δεύτερο το θέμα μου τι είναι να εξετάσουμε το α έως το ω πάλι όλη την πολιτική ασύλου. Εν πάση περιπτώσει, στα 10 λεπτά που έχω στη διάθεσή μου θα προσπαθήσω να κάνω κάποιες παρατηρήσεις τις οποίες διατυπώσαμε για το μελλοντικό αυτό σύστημα του Ευρωπαϊκού Ασύλου στον Οδυσσέα. Όπως και ο Φίλιπ Ντεμπρικέρ είπε στι αγωγικές του παρατηρήσεις, η πρώτη μου παρατήρηση είναι η εξή. Προφανώς θα πρέπει να κάνουμε μία επιλογή μεταξύ των θεμάτων που άπτονται της μεταρρύθμισης του παρόντος συστήματος και μια τρίτης φάσης, μια νέας φάσης. Σήμερα θα πρέπει λοιπόν να δούμε πώς μπορούμε να διορθώσουμε τις δηλειτουργίες που διαπιστώνουμε ότι πάνω στο παρόν σύστημα και να προσπαθήσουμε να προβλέψουμε και κάποια πράγματα πιο ριζοσπαστικά και πιο επαναστατικά για να διορθεί αυτή η κατάσταση. Και η εμπειρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση τι μας λέγει ότι ότι θα πρέπει να είμαστε πραγματιστές και η επανάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ο χρυσός κανόνας. Πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό, όντας συνεκτική και αποδοτική σε αυτή την πολιτική ασύλου. Θα ήθελα λοιπόν να σας προτείνω μια τριπλή προσέγγιση αν θέλετε όσον αφορά την δυνητική εξέλιξη της κοινή ευρωπαϊκής πολιτικής ασύλου. Μία πρώτα απ' όλα νομική, θεσμική, που θα προσπαθήσουμε περισσότερο να δούμε από ε, δικαιοδοτικής πλευράς τι σημαίνει. Λοιπόν, η νομική προσέγγιση προφανέστατα τίθεται με δύο τρόπους αυτή η προσέγγιση. Θα πρέπει πρώτα απ' όλα να σκεφτούμε τις δυνατότητες του άρθρου 18 του Θεμελιώδους Χάρτη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που προτείνει το δικαίωμα ασύλου έτσι όπως το εφαρμόσαμε μέχρι τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να το αναθεωρήσουμε. Για ποιο λόγο. Διότι εφ' το άρθρο 18 του χάρτη μας λέγει το δικαίωμα ασύλου είναι κάτι το οποίο εγγυάται βάσει τη Σύμβαση τη Γενέβη, τον τρόπο λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Γενέβη και τη Νέα Συνθήκη Λισαβόνα. Τι σημαίνει ότι ξεπερνά την απλή αναγνώριση και η λέξη εγγύηση και να εγγυηθούμε κάτι σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε κάτι περισσότερο από αυτά τα οποία να κάνουμε θεωρητικά όπω προβλεπόταν συνθήκη του Άμστερνταμ και του Μάστριχτ. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν πρώτα απ' όλα τι σημαίνει συγκεκριμένα αυτή η εγγύηση Τη τήρηση και του σεβασμού θεμελιώδου χάρτου ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πρόκειται αναμφίβολα για θεσμοθέτηση, αν θέλετε, του δικαιώματο ασύλου. Εφ' εξής, λοιπόν, βάσει του θεμελιώδους χάρτη, το δικαίωμα ασύλου ε, περιέχει και το κείμενο της Σύμβασης της Γενέβης και ό,τι αφορά τους πρόσφυγες. Δηλαδή έχουμε μία πράξη που μας επιτρέπει να εφαρμόσουμε πλήρως το δικαίωμα ασύλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, πάει πιο μακριά αυτό. Ίσως θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε. Ε, εφόσον λοιπόν το δικαίωμα ασύλου βασίζεται κυρίως στα κείμενα τα οποία το συνθέτουν, είναι προφανές ότι η, εφαρμοσι... η εφαρμοστικότητά του είναι κάτι το οποίο δεν είναι δύσκολο, μπορεί να ασκηθεί ε, βάσει των κειμένων που το συνθέτουν. Σύμβαση της Γενέβης, συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις διάφορες συνιστώσεις της, έτσι όπως ε, ε, καθορίζεται στον τρόπο λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται λοιπόν για μια σημαντική πρόοδο και δεν είναι προφανές ότι βάσει αυτής της πρόοδου δεν μπορούμε να καταλήξουμε σε κάποιες σε κάποια συμπεράσματα ότι όντως πρόκειται για εφαρμογή του δικαιώματος ασύλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πράγμα που μας προσφέρει, επαναλαμβάνω, η συνύπαρξη αυτών των κειμένων που προανέφερα. Δεύτερο ερωτηματικό, πάντα από νομικής πλευράς. Η ε, δυνατότητα προσχώρηση τη Σύμβαση τη Γενέβη. Πρόκειται για τεχνικό θέμα και πάω πολύ γρήγορα. Πολύ απλά, εδώ πρέπει να πω ότι άρχισε να συζητείται αυτό το θέμα διότι η Σουηδία και το πρόγραμμα δράσης για το δικαίωμα ασύλου αναφέρουν ρητά ότι πρέπει να δούμε ποιες είναι οι, δυνα... είναι οι δυνατότητες που προσφέρονται για την προσχώρηση στη Σύμβαση της Γενέβης. Κάτι τέτοιο είναι εφικτό. Είναι εφικτό για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα πρέπει να πω ότι έχει νομική προσωπικότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει αρμοδιότητε σε θέματα ασύλου, δεδομένου ότι θέλει να αναπτύξει κοινή πολιτική ασύλου, αλλά δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο καταρχήν η Ευρωπαϊκή Ένωση να προσχωρήσει στη Σύμβαση της Γενέβης. Μόνο που πρέπει να προσέξουμε το εξή. Τα πράγματα είναι πολύ πιο πολύπλοκο ότι φαίνονται. Το πεδίο εφαρμογή της Σύμβασης της Γενέβης ξεπερνά τις ε, αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε κάποιους τομείς υπάρχουν και ε, κοινέ αρμοδιότητες. Άρα έχουμε μια πολύπλοκη κατάσταση. Επίσης, εάν μελετήσει κανείς λίγο περισσότερο την ε, διάσταση της Σύμβασης Γενέβης, πρέπει να πούμε ότι εφαρμόζεται μόνο και δίνει πρόσβαση μόνο ίσως σε κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ένωσης βάσει πρωτοκόλων και συμφωνιών που προβλέπουν ότι ε, μπορεί να προσχωρήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με τα συμβαλόμενα μέρη επίσης στην ε, Σύμβαση της Γενέβης. Όλα αυτά εμπεριέχονται βεβαίως στην ε, έκθεση την οποία το δίκτυο Οδυσσέας θα δημοσιεύσει. Τώρα, θεσμική προσέγγιση. τι είναι η δυνατότητα που θα έχει αυτό το Ευρωπαϊκό Γραφείο για θέματα ασύλου. Προς το παρόν, για την, ε, τον οργανισμό αυτό υπάρχει μόνο μια συμφωνία, δεν μπορούμε να καταλήξουμε σε συμπεριμένοντα. Στα πλαίσια της ε, θεσμικής προσέγγισης μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν κάποια θέματα δυσλειτουργίας για τον οργανισμό αυτό που θα μπορούσαν να επιληθούν. Πρώτη δυσλειτουργία. Θα πρέπει να γίνει να γίνουν δεσμευτικές οι πράξεις αυτού του οργανισμού. Δεν είναι σοβαρό να λέμε σήμερα ότι αυτός ο οργανισμός θα συντονίζει τις ε, εθνικές πολιτικές και στο άρθρο 14 να λέμε ότι αυτά τα οποία κάνει αυτός ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός δεν είναι δεσμευτικές σε σχέση με τις αποφάσεις που παίρνει κάθε χώρα μέλος χωριστά. Κάποια στιγμή λοιπόν θα πρέπει αυτή την αντίφαση να τη διευθετήσουμε. Δεύτερον, θα πρέπει να μπορεί να γίνεται ε, ανάλυση της κάθε περίπτωσης βάση συγκεκριμένων παραδειγμάτων. Τρίτον, θα πρέπει να δούμε αν αυτός ο Ευρωπαϊκός Οργανισμό Ασύλου θα μπορέσει αύριο να μας επιτρέψει να επιλύσουμε κάποιες διαφορέ μεταξύ κρατών μελών και κατά τη διάρκεια τη μεταβατική περίοδου να κάνει και κάποια... να προτείνει κάποια διευθέτηση τέτοιου είδους διαφορών. Τώρα, Ας δούμε πώς μπορεί το θέμα της διαφοράς που μπορεί να υπάρξει αφορά τη διαδικασία που εφαρμόζεται σε περίπτωση προβλήματος που υπάρχει για το άσυλο. Εάν θεωρήσουμε ότι πρόκειται για ένα θεμελιώδες δικαίωμα, το άσυλο είναι ένα θεμελιώδες δικαίωμα και όχι μια απλή διαδικασία, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Άρα το η νομική διάσταση του όλου προβλήματος είναι σημαντική και θα πρέπει να τη λάβουμε υπόψη και σε αυτή την περίπτωση να ξεπεράσουμε κάποια μεγάλα εμπόδια. Ξέρετε ποιους εδιασμους εχουν έχουν κάποια κράτη-μέλη σε σχέση με τις αποφάσεις κάποιου ε, κοινοτικού δίκητη. Και σήμερα η διαχωριστική γραμμή μεταξύ των ε, προβλημάτων εθνικών διαφορών και κοινοτικών διαφορών πρέπει να πω ότι μπορούν να είναι πάρα πολύ μεγάλες. Ο εθνικός δικαστής κρίνει κατά την άποψή μου τις εθνικές αποφάσεις και τις υπόλοιπες τις κρίνει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Διότι ούτως ή άλλως το κράτος μέλος δεν παρέχει την ε, διεθνή προστασία, η Ευρωπαϊκή Ένωση την παρέχει. Άρα υπάρχει μία, ένα ορόσημο το οποίο είναι σαφώς καθορισμένο. Έτσι ο Ευρωπαίος δικαστής ποτέ δεν κυρώνει μία εθνική απόφαση. Μπορεί να ε, διαπιστώσει ότι είναι σωστή, ότι μπορεί να ενδέχεται έφαση, αλλά δεν μπορεί να την ε, ακυρώσει ή να την ε, ανακαλέσει. Μόνο ένας εθνικός δικαστής μπορεί να το κάνει. Θα πρέπει λοιπόν πρώτα απ' όλα να εκλογικεύσουμε κάπως τα πράγματα για να προχωρήσουμε. Τι σημαίνει αυτό. Ότι αν η εναρμόνιση της πολιτικής ασύλου είναι κάτι το οποίο είναι από κανονιστικής πλευράς αποδεκτό, δεν είναι αποδεκτή από άποψης δικαιοδοσίας. διότι ανάλογα με το που βρίσκεται ο πρόσφυγας και ανάλογα μπροστά σε ποιες εθνικές αρχές ζητά άσυλο, του εφαρμόζεται διαφορετικό εθνικό δίκαιο. Θα πρέπει λοιπόν αυτό να το λάβουμε υπόψη και για να είμαστε ε, δίκαιοι και αποδοτικοί θα πρέπει να δούμε πώς θα ιεραρχήσουμε τις προτεραιότητες για να κάνουμε κάτι το αποδοτικό. Πριν ε, να ε, προσφέρει λοιπόν τη δυνατότητα προσφυγής στους ε, ετούντες άσυλο θα πρέπει να δούμε πρωτογενώς πώς θα μπορέσουμε να εναρμονίσουμε τις διαδικασίες που προβλέπεται τη χορήγηση ασύλου σε όλα τα δίκαια. Και μέσω αυτού του οργανισμού για τη χορήγηση ασύλου θα πρέπει να προσπαθήσουμε να ε, υποχρεώσουμε κατά κάποιο τρόπο τα κράτη-μέλη να ακολουθούν παρεμφερείς διαδικασίες. Καταρχάς ελέγχθη ότι κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατό. Αλλά θα πρέπει να δούμε το εξή. Αυτός ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σύλλου, τα πλαίσια της διακριτική ευχέρειας του καθενός θα πρέπει να μπορεί να δημιουργήσει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο ο καθένας θα μπορεί να κινηθεί. Α πάρουμε ένα άλλο τομέα, τον τομέα τη ανταγωνιστικότητα, του ανταγωνισμού και ε, των γενικών γραμμών και του πλαισίου που υπάρχει λέει το Ευρωπαϊκό ε, Δικαστήριο, αν θέλει κάποιος να υπερβεί τα πλαίσια, θα πρέπει να το αιτιολογήσει. Δηλαδή, σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση, εάν κάποιο κράτος θέλει να υπερβεί τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές που θα τεθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πρέπει να αιτιολογήσει τα, ε, τις πράξεις του. Πράγμα που θα επιτρέψει αφενός βασιζόμενοι στη συνθήκη της Λισαβόνας που μας επιτρέπει να έχουμε προσφυγή βάση πράξεων κάποιων οργανισμών, πρώτα απ' όλα να ελέγχουμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί και αποφασίζει αυτός ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασύλου, διότι μπορεί ενδεχομένως αυτός ο οργανισμός να δώσει κάποιε κατευθύνσεις γραμμές εντελώ αντίθετε προ τη συνθήκη της Λισαβόνας. Δεύτερον, γιατί εμείς δεν θα χρησιμοποιούμε την δυνατότητα που μας δίνει η συνθήκη του Άμστερνταμ. Δηλαδή, προ όφελο του νόμου να κάνουμε προσφυγή εάν υπάρχει προφανής αντινομία μεταξύ των γενικών γραμμών και της πολιτική ενό κράτου, να δούμε ποιε είναι οι απαιτήσει του ε, κοινοτικού δικαίου. Στην κατάσταση στο Ιράκ, Φερρυπίν, είδαμε ότι για κάποιες χώρες η κατάσταση θεωρείται ως μία κατάσταση ακραίας βίας, άρα αιτιολογεί κάποιες πράξεις από κάτι μέλη, για άλλες χώρες πρόκειται για μία γενικότερη κατάσταση πιο χαλαρή και για μία μοιραία εξέλιξη. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε τα πράγματα χωρίς διασύνη δεδομένου ότι είναι πάρα πολύ πολύπλοκο το όλο θέμα και θέλουμε ότι κάνουμε να το κάνουμε με πλήρη σαφήνεια. Ευχαριστώ. Thank you, uh, I will now open the... Ευχαριστούμε καθηγητά. Να ξεκινήσουμε τώρα την συζήτηση. Θα ζητήσω από όσους θέλετε να θέσετε ερώτημα να εκδηλώσετε άμεσα τον ενδιαφέρον σας. I understand that at one point... Ε, ότι κάποια ερωτήματα έχουν ήδη τεθεί αλλά ε, ίσως θέλουν κάποιοι να παρέμβουν. Ποιος θα σπάει στον πάγο. Ο κίνδυνος είναι να συνεχίσω να ομιλώ για κάνα μισάωρο. I ε, Καθηγητά Λαμπάιλ, Σημειώσατε ενδεχομένω τα ερωτήματα που τέθηκαν στι πρώτε φάσει τη συζήτηση. Μήπω να σχολιάζετε αυτά τα σημεία ευθύ αμέσω ότου άλλοι συνάδελφοι έρθουν με άλλα ερωτήματα. Νομίζω το βασικό θέμα που τέθηκε προηγουμένω αφορούσε τι προοπτικές που προσφέρονται από την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Συνθήκη για, τις... για τα δικαιώματα του ανθρώπου. Το θέμα εδώ είναι αν πραγματικά πρόκειται για επανάσταση ή όχι. Νομίζω ότι κατά πρώτον καλό είναι να θυμόμαστε ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και επειδή η Ευρωπαϊκή αυτή σύμβαση δεν εγγυάται το δικαίωμα ασύλου, ο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δεν είναι ο ευρωπαικο δικαστηριο ανθρωπινων δικαιωματων δεν ειναι ο για αυτές τις περιπτώσεις. Παρεμβαίνει για να προστατεύσει δικαιώματα που τα ίδια διασφαλίζονται από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ιδίως το άρθρο 3, απάνθρωπη μεταχείριση ή <clears throat> κακομεταχείριση, ε, παράνομη επαναπρόθεση ή αρμονικός οικογενειακός βίος. Τώρα το παράδοξο που δημιουργείται, να υπάρξει προσχώρηση δηλαδή και να παρεμβαίνει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στο περιθώριο των Ευρωπαϊκών Πλουτών, αυτό σημαίνει ότι ο Ευρωπαίος Δικαστής θα ελέγχει την επικουρική προστασία, αυτή το άρθρο 3. Ενώ το θεμελιώδες δικαίωμα των προσφύγων που προκύπτει από τη Σύμβαση, από τη σύμβαση της Γενέβης δεν θα προστατεύεται από κάποιο δικαστή. Ποιο συνεπές λοιπόν θα ήταν να έχουμε περισσότερη δικαιοδότηση από ό,τι σήμερα. Δηλαδή, εντό τη ε, κοινή πολιτική ασύλου, οι δύο πτυχέ, επικουρική προστασία και βασική προστασία, να ελέγχονται από έναν και μόνο δικαστή. Αυτό είναι η πρώτη μου παρατήρηση. Η δεύτερη είναι ότι ο έλεγχο που γίνεται από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων επιτρέπει να σκεφτεί κανεί ότι μετά την προσχώρηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι επικουρικό έλεγχο. Και αυτό γίνεται όλο και πιο ξεκάθαρο <clears throat> με αυτή την προσχώρηση. Και εδώ μιλάμε για συγκεκριμένε υποθέσει, περιπτώσει, όχι για τι αρχέ. Δεν θα ελέγχει την νομιμότητα μια πολιτική, θα υπάρχει έλεγχο επί συγκεκριμένων περιπτώσεων. Αυτέ προκύπτουν καθημερινά με την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και πάλι λοιπόν, η άνοδο τη εξουσία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δεν πρέπει να μα επιτρέψει να σκεφτόμαστε ότι θα καταλήξουμε σε αποτέλεσμα ανάλογο με αυτό που θα έχει πλήρη ανάληψη ελευθεριών από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο τη Ευρωπαϊκή Ένωση των θεμάτων αυτών. Όλα λοιπόν συνηγορούν υπέρ του Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει τι ευθύνε τη. Είτε με τρόπο γενικό είτε με τρόπο εξειδικευμένο. Ό,τι και αν επιλέξουμε βλέπετε ότι η επιλογή ενό ειδικού δικαστηρίου περί θεμάτων ασύλου είναι, αποκλείεται για την ώρα. Διότι υπάρχουν ανάλογες ρήτε στη συνθήκη και επειδή θέλαμε τις στη μελέτη που κάναμε να χρησιμοποιήσουμε τις αρχές της συνθήκης που ισχύει. Δεν μπορούμε να υποθέτουμε ότι θα μετατρέπεται και θα αλλάζει η συνθήκη κάθε πρωί. Το ειδικό δικαστήριο λοιπόν περιθυμάτων ασύλου φαίνεται να είναι μια προοπτική πολύ απίθανη, σχεδόν ακατόρθωτη. Θα πρέπει λοιπόν μαζί με το ευρωπαϊκό, μαζί με τα προκαταρτικά με τα προδικαστικά μάλλον ερωτήματα, με τις αιτήσει για κύρωση, τι προσφυγές, τις ανασταλτικέ, όλες αυτές οι υποθέσει να μπορούσαν να εξετάζονται από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, διότι ο πραγματικό δικαστή σε κάθε περίπτωση για τα θέματα ασύλου είναι ο εθνικό δικαστή πριν φτάσουν αυτά τα θέματα στον Ευρωπαϊκό Δικαστή. Θα έλεγα, πιστεύω, ότι το ΔΕΚ, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, στο μέλλον πολύ πιο έντονα με θέματα μετανάστευσης ε, και ασύλου θα επομίζεται. Και δεν είμαι βέβαιος αν αυτή η διαδικασία που έχουμε θα είναι η σκόπιμη και η πιο εύλογη σε αυτή τη διεργασία επαρκώς γοργά και με επαρκή σαφήνεια να μπορούμε να καταλήξουμε στην ερμηνεία του ευρωπαϊκού δικαίου για το άσυλο και τη μετανάστευση. Γι' αυτό και η σκέψη μου, ο προβληματισμός μου, αν δεν θα έπρεπε να δημιουργήσουμε μια διαδικασία που κάπως να είναι συγκρίσιμη με τις διαβουλευτικές συμβουλευτικές ε, επιτροπές ε, ή και να δίνεται η δυνατότητα στο δικαστήριο ως με το μέσο αμίκους κούριε του ε, βοηθού του δικαστηρίου να ε, επικουρεί το δικαστήριο για θέματα μετανάστευσης και ασύλου και να δίνεται η δυνατότητα να ακολουθεί το δικαστήριο αυτές τις γνωμοδοτήσεις ή όχι. Αυτή η Επιτροπή θα, θα συνετίθετο από ομάδα ατόμων που πολύ πιο εξειδικευμένα και που πολύ πιο γοργά θα μπορούσε να αποφασίζει για τέτοια θέματα και που θα μπορούσε να έχει μια μεγαλύτερη επισκόπηση για την εμβέλεια των θεμάτων αυτών. Ένα κάποιο πρόβλημα βλέπω και βρίσκω και αυτό επισημάθηκε πιο πριν στο εξή θέμα, στο ότι οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου είναι αναπερίπτωση νομολογίες όμως ερμηνεύονται ή συλλέγονται και εκτίθενται με γενικό τρόπο στην πρακτική ε, νομική ζωή των κρατών μελών. Και από αυτό απορρέει μια πληθώρα δυσκολιών. Έχουμε οδηγίες για τα κράτη-μέλη από, ε, τοποθετη... από γνωμοδοτήσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου ή νομολογίες. Και από αυτά δημιουργούνται σοβαρές ε, δυσκολίες διότι δεν έχει σωστά αναγνωριστεί ότι τα δικαστήρια έχουν μια διαφορετική ε, εξουσία και καθήκον από τον Ευρωπαίο νομοθέτη. Ο Ευρωπαίος νομοθέτη πρέπει γενικά να θέτει τις αρχές που θα ισχύουν στο μέλλον σε ένα νομικό πλαίσιο. Τα δικαστήρια αποφασίζουν περιπτώσεις και συγκεκριμένα θέματα και δεν μπορεί κανείς από μια νομολογία του δικαστηρίου, ενός δικαστηρίου να μπορεί κανείς να ε, καταλήγει σε νομοθετικές ρυθμίσεις. Ευχαριστώ partage évidemment euh, l'opinion de Συμμερίζουμε την άποψη του κ. Χάιλμπρονερ. Απλώς δύο διαπιστώσεις, μία πολιτικού χαρακτήρα. Το δικαστήριο θα έλεγα ότι ζηλεύει ιδιαίτερα για αυτές τις ε, αρμοδιότητες. Εδώ και κάποια χρόνια μιλάμε για εξειδίκευση, μιλάμε για συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, ώστε να απαλλαγεί από κάποιες από τις αρμοδιότητές της, αλλά τελικά τίποτε δεν γίνεται. Η διοργάνωση εξέταση και επίλυση διαφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει αντάξει τα τελευταία 30-40 χρόνια. Παρά την εμφάνιση του πρωτοβάθμιου, του πρωτοδικίου μάλλον, έτσι έχουν, μπορούμε να δούμε τα πράγματα για την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπάρχει ειδικό πρωτοδικείο για τα ζητήματα που εξετάζει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Αυτό είναι το πρώτο στοιχείο. Έπειτα, για τα θέματα του ασύλου υπήρξαν πολλές ε, φαντασιο, ονειροφαντασίες και σχέδια, αλλά κανένα τεκμηριωμένο γεγονός. Πρέπει να δούμε λοιπόν αν η ροή των, υποθέσεων που θα φτάσουν ενώπιον αυτών των δικαστών είναι αρκετά ε, σοβαρή, ώστε να δικαιολογεί τη δημιουργία τέτοιου οργάνου. Όταν το πρωτοσυζητήσαμε, ε, πολλά κράτη μεταξύ των οποίων και το δικό μου φοβήθηκαν ότι 300.000 αιτήσει ασύλου θα φτάσουν στα χέρια ενό δικαστή ενδεχομένω στο Λουξεμβούργο, εφόσον δημιουργεί το. Αλλά αυτά βάσει του Άμστερνταμ. Και στι πρώτε διαπραγματεύσει για αυτή τη συνθήκη είπαν ότι θα υπάρχει κυκλοφοριακή συμφόρηση στη δικαιοδοσία, εάν γίνει κάτι τέτοιο. Τώρα δεν μπορούμε να προβλέψουμε αν θα υπάρξουν δυακόσες, 200, δύο 2.000, ένα εκατομμύριο αιτήσει. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Θα πρέπει όμω να είμαστε σε θέση να εξετάσουμε και το φόρτο που θα αναλογεί σε ένα τέτοιο δικαστήριο. Και τρίτη παρατήρηση είναι αυτό που είπε προηγουμένω, Σκάι. Το έχουμε συζητήσει και με τον κύριο Ζωμότ. Νομίζω ότι υποτιμούμε εδώ τη σημασία τη ταχύτητα, τη ταχύ επίλυση τέτοιων ε, υποθέσεων. Προηγουμένω μιλήσαμε για την κράτηση προσώπων. Αλλά αυτό πολλές φορές έχει να κάνει και με την αδυναμία μας να δώσουμε μια αξιόπιστη και ταχεία απάντηση στο εξή. Ο ετών αξίζει ή όχι να έχει προστασία δικαιολογημένη. Όλοι λοιπόν οι μηχανισμοί που σήμερα λειτουργούν και όλες οι οι αλληλοσυγχαντισμοί που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν επιτρέπουν αρκετά άμεσα να απαντήσουμε στην αίτηση ενό κράτου ή στο αίτημα μια εθνική δικαιοδοσία που θέλει μέσα σε τρει μέρε να έχει απάντηση στο ερώτημα που θέτει. Άρα πιθανώ εδώ για τα θέματα του ασύλου υπάρχει ανάγκη εξειδίκευση. Κυρία Λάμπερτ, να θέσω ένα ερώτημα για το τι πιστεύετε ότι θα μπορούσε να λάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως ρόλο μέσα σε όλα αυτά. Διότι μέρος του ρόλου της είναι η παρακολούθηση και τα λοιπά. Αλλά το είδαμε και σε σχέση με τις δικές μας αρμοδιότητες στο κοινωνικό τομέα. Εάν υπάρχουν προβλήματα στην υλοποίηση, τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να, να διευκολύνει την υλοποίηση ενό συγκεκριμένου νομοθετήματο. Συνήθως καταλήγει σε κατευθυντήριε γραμμέ. Και μία από τι βασικέ αρμοδιότητε που ανατέθηκε στο γραφείο για το άσυλο είναι είναι η εξέταση στοιχείων που ελέγχονται από το γραφείο ενώ παρακολουθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πού νομίζετε λοιπόν ότι εντάσσεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε όλο αυτό το τοπίο. Ήδη το γεγονός ότι δυσκολεύομαι να σας απαντήσω είναι ένα είδος απάντησης. Εάν ε, ερμηνεύατε την απάντησή μου ήδη, θα καταλαβαίνετε ότι δεν εντάσσεται σε όλο αυτό το πλαίσιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Αναντήρητα σήμερα, Υπάρχει μια φυγή των θεσμικών οργάνων από την εξέταση αυτών των προβλημάτων. Προσπαθούν να απαλλαγούν από κάποιες δυσκολίες. Και επιτρέψτε μου να χρησιμοποιήσω εδώ μια έκφραση ιδιαίτερα γαλλική. Προσπαθούν να δώσουν τα κάστανα τα καυτά στον γειτονά του. Για να μην καούν οι ίδιοι. Υπάρχουν λοιπόν διάφοροι μηχανισμοί που λειτουργούν παράλληλα, χωρίς κανείς να διερωτάται για το πώς ορισμένοι μηχανισμοί υλοποιούνται πραγματικά και πώς ελέγχονται. Σήμερα το γραφείο για το άσυλο μπορεί να είναι μια τέλεια ευκαιρία για τη δημιουργία μιας κοινή πολιτικής ασύλου και για να είναι πολιτική αυτή σοβαρή. Όμως ποιο σήμερα θα προσπαθήσει να παρακολουθήσει το γραφείο αυτό και να εξετάσει αν λειτουργεί συνεκτικά και αποτελεσματικά. Δεν είχα το χρόνο να το πω προηγουμένω. Υπάρχουν δυνατότητε. Τι προβλέπουν τα κείμενα όπω ισχύουν σήμερα για το Ευρωπαϊκό Γραφείο Ασύλου. Λόγω χάρη η δυνατότητα των ομάδων εργασιών να κατονομάζουν δικαστέ. Νομίζω ότι η ερμηνεία των ε, ρητρών για το άσυλο από την πλευρά ενό δικαστή δεν θα είναι ίδια ποτέ με ενό δημοσίου υπαλλήλου ή ενό υπευθύνου που δουλεύει στο οργανισμό αυτό. Η σύνθεση η συνθεση λοιπόν του οργανισμού για το άσυλο μπορεί να επιτρέψει να δημιουργηθούν ε, σχέσεις δυναμικές καθόλου. Ε, το να προβλεφθεί μια προσέγγιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων ρεαλιστική που να λαμβάνει υπόψη τις εθνικές δυσκολίες, τις ευαισθησίες των κρατών μελών, την ε, βούληση που έχουν οι εθνικές δικαιοδοσίες να διατηρήσουν κάποια δικαιώματα, το δικαίωμα της πρωτοβουλίας των ε, κυρίαρχων κρατών. Όλα αυτά είναι το πλαίσιο της πραγματικότητας που πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Όμως, βάσει του πολιτικού ορθού σήμερα, αποφεύγουμε τα ερωτήματα αυτά και υπεκφεύγουμε Γι' αυτό κάποια συγκεκριμένα άτομα, οι άνθρωποι οι ίδιοι, είναι τα θύματα αυτής της κατάστασης. Κάτι που πραγματικά είναι απάνθρωπο. Ε, Ευχαριστούμε. Υπάρχουν άλλοι που ζητούν να παρέμβουν, παρακαλώ. Αν δεν ζητεί κανείς να παρέμβει, τότε θα ολοκληρώσουμε την εκδήλωσή μας. Ο καθηγητής δεν θα ήθελε να κάνει μια σύντομη παρατήρηση για να κλείσει η συνεδρίασή μας. Έχετε τον λόγο, καθηγητά. Uh, Φυσικά όχι μια καταληκτική ε, παρατήρηση αλλά μια πρακτική υφής πληροφορία. Όπως ίσως ε, κατανοήσατε η μελέτη μας δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Ολοκληρώνουμε σταδιακά τη μελέτη μας και είναι δύσκολο το εγχείρημα και είναι και ευρύτατο το θέμα και έχουμε κάθε εβδομάδα σχεδόν νέα έγγραφα, νέα στοιχεία, νέες πληροφορίες που πρέπει να εντάξουμε στη μελέτη μας. Παρ' όλα αυτά όμως σιγά σιγά ολοκληρώνεται και θα υπάρξει και συζήτηση φυσικά με τις αρχές, ε, με τη διοίκηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επ' αυτής της μελέτης ώστε να ολοκληρωθεί η μελέτη αυτή ίσως και την επόμενη εβδομάδα. Μετά θα δημοσιευθεί αρκετά σύντομα αυτό το οποίο δεν γνωρίζω φυσικά είναι αν αυτό θα γίνει πριν ή μετά τις θερινές διακοπές. Όμως είναι σχεδόν βέβαιο ότι η μελέτη αυτή θα είναι διαθέσιμη σύντομα και θα βρείτε επίσης και σε αυτή τη μελέτη πολλά περισσότερα στοιχεία από αυτά τα οποία ακούσατε εδώ σήμερα. Διότι εδώ επιλέξαμε επιλεκτικά 6-7 ζητήματα ή θέματα. Στη μελέτη έχουμε πολλά περισσότερα και σε βάθος τα εξετάζουμε. Τα θέματα αξιολόγησης, αποτίμησης, τα θέματα του κεκτημένου, τα θέματα το θέμα του μέλλοντος ε, που θα έχει το ευρωπαϊκό σύστημα Σύλλου στο μέλλον μακροπρόθεσμα. Αυτό ελπίζω ότι θα ανοίξει την όρεξή σας να διαβάσετε τη μελέτη αυτή υστερότερα και ότι θα είναι χρήσιμη σε εσά. Και θα δούμε αν θα μπορέσουμε υστερότερα να κάνουμε και μία ακόμα παρουσίαση επί του πλήρου κειμένου και εύρου τη έκθεση. Σα ευχαριστώ που είσαστε παρόντε εδώ και ευχαριστώ ιδιαίτερα την Ευρωβουλή που μα καλωσόρισε και μα έδωσε αυτή τη δυνατότητα. Σα ευχαριστούμε κύριε καθηγητά, λέει κύριο Μπούσετηρ. Ευχαριστώ επίση ε, και τον καθηγητή ε, Βαλ για την παρουσίαση σε, αυτή την, ε, σε αυτό το τμήμα τη συνεδρίαση και όλου του άλλου που παρενέβησαν σήμερα σας φιλοξενούμενοι. Σας, σας ευχαριστούμε εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς επίσης ε, ευχαριστούμε και τους συναδέλφους από τα Εθνικά Κοινοβούλια που ήταν παρόντα εδώ σήμερα ως μέλη, καθώς επίσης ε, και του δικτύου. Σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας, την υπομονή σας, την ε, ενεργό συμμετοχή σας και έτσι λίγη συνεδρίασή